Dear colleagues, dear guests, I think that we... Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν λοιπόν καλωσορίσω και συστήσω τους συναδέλφους και καλεσμένους μας, θα ήθελα να ξεκινήσω με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξής μας, όπου υπάρχει μια αλλαγή ε, σχετικά με το σημείο 9, το οποίο αναβάλλεται μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, οπότε θα υπάρχουν ε, και όλοι οι γλωσσικοί συνδυασμοί. Δεν βλέπω αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Περνάμε τώρα στο δεύτερο σημείο της σημερινής διάταξης. Δεν έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις όσον αφορά την ε, έγκριση λοιπόν ε, των ε, παρακτικών σχετικά με τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου, 28 Ιανουαρίου, της 1ης Φεβρουαρίου, καθώς επίσης και τη συνεδρίαση των 17 και 18 Φεβρουαρίου. Θεωρούνται λοιπόν ότι γίνονται δεκτές, έτσι λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε στο σημείο 4, το οποίο αφορά την ακρόαση για την ε, προστασία των ευπαθών ενηλίκων. Και θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους ε, ομιλητές μας, αρχικά με τον κύριο Ντομένικο Νταμαστέλη, ο οποίος είναι ε, Ιταλός ε, συμβολιογράφος, την κυρία ε, Άννε και Φρένεγκορο, η οποία είναι νομική σύμβουλος σχετικά με τη διεθνή διαχείριση ακινήτων. Θα περάσω στον κύριο Φρίμστον, δικηγόρο, καθώς επίσης και τον κύριο Ρέγκα, ο οποίος είναι συμβολιογράφος από την Γαλλία ε, και ελπίζω να έχουμε και τον ε, κύριο ε, Φιλίπ Λεκάφ μαζί μας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του οργανισμού για, τον ιδιωτικό, για το ιδιωτικό, διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Θα περάσουμε τώρα στις νομικές υποθέσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως, δίνοντας το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, που είναι ο κύριος Νταμαστέλη. Συγγνώμη, ελπίζω να έχω προφέρει σωστά το όνομά σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους όσους θα πάρουν το λόγο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που συμμετέχω για δεύτερη φορά σε συνεδρίασή σας. Η πρώτη φορά ήταν πριν 10 χρόνια σχετικά με την κληρονομία σε περίπτωση θανάτου. Η διαδικασία που είχε τότε ξεκινήσει οδήγησε στην υιοθέτηση της, του κανονισμού 650 ε, του 12 που είναι από τις πιο αν θέλετε φιλόδοξες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ιδιωτικό διεθνές. Νομίζω ότι και στον, τον τομέα στον οποίο σήμερα καλούμε να κινηθούμε να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Η ανάγκη να μην μακρηγορήσω. Με εμποδίζει από το να υποδείξω λεπτομερώς θα έλεγα τους λόγους για τους οποίους ε, καθίστανται απαραίτητες αν όχι εύθετες οι παρεμβάσεις του Ευρωπαίου ε, νομοθέτη στον τομέα της προστασίας των ευάλωτων ε, ανηλίκων. Γι' αυτό ακριβώς η απουσία κοινών κανόνων μερικές φορές ε, ε, οδηγεί στον καθορισμό του ε, αρμόδιου δικαστή για τα μέτρα προστασίας του προσώπου και της περιουσίας του. Στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου σε κάθε περίπτωση και στην εγγύηση κυκλοφορίας των αποφάσεων αυτών στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Χώρου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των συγκεκριμένων προσώπων αυτών από τις πρωτογενείς πηγές δικαίου της Ένωσης. Σε αυτές τις παρατηρήσεις να προσθέσω δύο επιπλέον, οι οποίες θα με οδηγήσουν και στην παρουσίαση του θέματος του κεντρικού της παρέμβασής μου. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην ηλικιώδη αύξηση του αριθμού των ανηλίκων που σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα βρεθούν τα επόμενα χρόνια λόγω του προχωρημένου της ηλικίας ή λόγω αναπηριών παθολογικών ή ψυχολογικών στην αδυναμία να φροντίσουν τα συμφέροντά τους προσωπικά. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προσώπων αυτών θα είναι κάτοικος του κρατών μελών, των εδαφών των κρατών μελών, όπου περισσότερο από άλλες περιοχές του κόσμου οι συνθήκες ζωής και ένα καλό επίπεδο κοινωνικής αρρωγής θα διασφαλίσουν ε, μια μακρό θα έλεγα ένα μακρύ προσδόκιμο ζωής. Η δεύτερη παρατήρηση ε, αφορά την επαγγελματική μου εμπειρία. Πολλοί από αυτή την κατηγορία απευθύνονται σε μένα όπως και σε άλλους Ιταλούς συναδέλφους και συναδέλφους άλλων χωρών έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες μιας επερχόμενης στο μέλλον αναπηρίας όταν ακριβώς ε, δεν μπορούν να την αποφύγουν βέβαια και υφίστανται μια άρνηση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων τους λόγω του περιεχομένου της ισχύουσας νομοθεσίας. Πρέπει να παρατηρήσουμε επίσης ότι στις περισσότερες χώρες η προστασία των ε, ενηλίκων των ε, ευάλωτων ρυθμίζεται με βασικούς κανόνες που επιτρέπουν μόνο εκ των υστέρων την παρέμβαση της νομοθεσίας αφού έχει προηγηθεί προσφυγή σε ειδικό ιατρό. Η προστασία αυτή επίσης επαφίεται και στους δικαστές οι οποίοι ορίζουν μερικές φορές έναν κηδεμόνα και εκδίδουν τις απαραίτητες άδειες για τη διαχείριση της περιουσίας του αναπήρου έτσι ώστε ε, να υπάρχει τακτική πρόσοδος για την επιβίωσή του και επίσης ε, να μπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις ε, δημοσιοποίησης των οικονομικών του δραστηριοτήτων. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικούς τρόπους ορισμού αυτών που φροντίζει και εκπροσωπεί το συγκεκριμένο πρόσωπο λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες αλλά και τα προγράμματα ίσως τα οποία μπορεί να έχει και να θέλει να εφαρμόσει στο μέλλον το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αναφέρομαι στο Vorsorgevollmacht που προβλέπεται από το γερμανικό δίκαιο, στο Lasting Power of Attorney το οποίο ε, ισχύει στην Αγγλία από το 2005 και στην Ιουλία, όπως επίσης και το Mandat de Protection Future σύμφωνα με τα άρθρα 477 του Γαλλικού Αστικού Κώδικα. Τέτοια μέσα θεωρούνται συμφωνίες ανάμεσα στον εντολέα και τον εντολοδόχο ή και σαν μονομερείς δηλώσεις ε, του εντολέα και ταυτόχρονα συνοδεύονται από μία σειρά άλλων στοιχείων αφήνουν στον εντολέα τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ακριβώς το εύρος του accertata da un terzo, non escludono l'intervento del giudice in funzione di controllo della... Το εύρος της εξουσιοδότησης... In dubbio che il legislatore europeo deve guardare a strumenti di... Ok, και ταυτόχρονα τέτοιου είδους μέσα θα πρέπει θα έλεγα να ερευνηθούν προσεκτικά. Εξυπηρετούν ένα διπλό στόχο, ο οποίος είναι συμβατός με το δίκαιο της Ένωσης. Πρώτον, ε, γίνεται προσπάθεια αποφυγής περιορισμού ε, της ε, παρέμβασης της δικαστικής εξουσίας και διευκολύνουν την διοικητική λειτουργία θα έλεγα σε επίπεδο δικαιονομικό. Ταυτόχρονα δευτερευόντως επιτρέπουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο να επιλέξει ε, τα ε, υποκείμενα τα οποία θα ασχοληθούν με την φροντίδα του ή στο μέλλον και ταυτόχρονα θα δώσουν εγγυήσει για την αυτοδιάθεση του ανθρωπίνου προσώπου ακόμα και σε μια ευαίσθητη στιγμή της ζωής του θα διασφαλίσουν την κυδαιμονία με αποτελεσματικό τρόπο γιατί οι διαδικασίες μερικές φορές οι δικαστικές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν η επικύρωση ή και η συμμετοχή στη σύμβαση της ΆΙΑ για την προστασία των ενηλίκων της 13ης Ιανουαρίου του 2000 μπορεί να ευνοήσει ε, την εφαρμογή των μέσων τα οποία περιγράψαμε. Η Συμφωνία της Χάγης λοιπόν λαμβάνει υπόψη από τη μία τα μέσα αυτά, ιδιαίτερα το άρθρο 15, εντοπίζει το νόμο ο οποίος εφαρμόζεται στη συμφωνία αυτή από την μονομερή ενέργεια ενός ενηλίκου προς ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα τον εκπροσωπεί έτσι αποφασίζει. Είναι αρκετά ελαστική η περιγραφή αυτής της πράξης σχετικά με και τις προβλέψεις κύρωσης της συγκεκριμένης ρύθμισης από πλευράς των κρατών μελών. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης μιας εναλλακτικής λύσης σύμφωνα με τη νομική ρύθμιση της συγκεκριμένης χώρας ή μιας διαφορετικής χώρας ανάλογα με το τόπο στον οποίο βρίσκεται η περιουσία. Παρ' όλα αυτά η σύμβαση δεν διασφαλίζει ε, πράξεις τέτοιου είδους να κυκλοφορούν χωρίς εμπόδια και να ισχύουν σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προέρχεται γιατί από το ότι το τέταρτο κεφάλαιο της σύμβασης καθορίζει την αναγνώριση και την εφαρμογή της συμφωνίας μόνο για τα μέτρα προστασίας του ενηλίκου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του άρθρου 22, το οποίο από τη μία αναφέρεται στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τις αρχές ενός συγκεκριμένου κράτους που είναι αρμόδιες επί τη βάση της νομικής ρύθμισης για τέτοιου είδους ενέργειες και από την άλλη περιλαμβάνει ένα κατάλογο ε, αιτιών ε, που δικαιολογούν ίσως τη μη αναγνώριση μιας τέτοιας διαδικασίας. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί ίσως να επιληθούν μέσω και του άρθρου 38 της Σύμβασης. Εξάλλου τέτοιου είδους ε, εγγυητικά συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να ισχύσουν μόνο εφόσον οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της σύμβασης ε, καλύπτουν την συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογα με την επιλογή της νομικής διαδικασίας και ανάλογα με τον νόμο ο οποίος εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο κράτος. Πρέπει να πούμε επίσης ότι μια τέτοια δευτέρου επίπεδου διοικητική διαδικασία ε, δεν είναι πάντα απαραίτητη να ισχύει και στις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και στην περίπτωση που η εντολή παίρνει τη μορφή ε, μια συμβολιογραφικής πράξης όπως Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία και στην περίπτωση που ενσωματώνεται μια τέτοια πράξη σε μια ευρύτερη πράξη όπως στην Αγγλία και στην Ουαλία όπου μια, ένα αντίγραφο πιστοποιημένο της εντολής δημοσιεύεται στο Public Guardian μετά από την καταγραφή. Και έτσι τέτοιου είδους πράξεις θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και από τα άλλα κράτη-μέλη. Ένα χρήσιμο τέτοιο πρότυπο, απο, πρότυπο αποτελεί το άρθρο 59 και το άρθρο 60 του κανονισμού 65212 για τη κληρονομιά. Ένα άλλο πρόβλημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι η σύμβαση αυτή δεν καθορίζει τις διαδικασίες για την ε, κυκλοφορία αυτού του είδου του πιστοποιητικού. Η ελάχιστη χαμηλή εμπιστοσύνη που έχουν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της σύμβασης μαρτυρείται από το ότι κανένα από τα κράτη που εφαρμόζουν την σύμβαση αυτή ε, δεν ε, έχουν δηλώσει στην διάσκεψη που την ορίζει το όνομα της αρμόδιας αρχής για την έκδοση των πιστοποιητικών εγγράφων. Αλλά το βασικό πρόβλημα της σύμβασης είναι ότι δεν προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την έκδοση της εντολής υποεξέταση. Τέτοιου είδους όρια δεν υπάρχουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 81 του της συνθήκης λειτουργίας προβλέπει σαν μέσο δικαστικής συνεργασίας και την υιοθεσία μέτρων που έχουν σαν στόχο την γυτνίαση των νομοθεσιών των κρατών μελών. Στα πλαίσια μιας τέτοιας προοπτικής, εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει στην εναρμόνιση των μέτρων, εάν αρνηθεί να προχωρήσει στην εναρμόνιση αυτή σε σχέση με ένα αυτόνομο διοικητικό μέσο, και εκεί γίνεται υποχρεωτική η επικύρωση ουσιαστικά ή μάλλον αρκείται στην επικύρωση από πλευράς των κρατών μελών της Σύμβασης της Χάγης, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει ανάγκη για, μια, για ένα συμπληρωματικό κανονισμό, ο οποίος να καλύπτει τις βασικές ανησυχίες της παρέμβασής μου. Γνώμη μου είναι ότι αυτός ο κανονισμός θα ήταν χρήσιμος και θα πρέπει να καλύψει το θέμα της εισαγωγής στις νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών που υπάρχουν ελλείψεις, ανάμεσα και στα άλλα άμεσα εφαρμόσιμα μέσα μέσω του κανονισμού σαν παράδειγμα και ένα πρότυπο ενός ε, μιας εντολής ε, η οποία προβλέπει την δυνατότητα για κάποιον ενήλικα και ικανό να παίρνει αποφάσεις να δώσει την δυνατότητα σε ένα ή και σε περισσότερα πρόσωπα να τον εκπροσωπήσουν και να ε, εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά του ε, εφόσον ο ίδιος καταστεί ανίκανος, που προβλέπουν επίσης τις διαδικασίες βεβαίωσης της αναπηρίας, δίδοντας στην εντολή την δυνατότητα να ορίσει άμεσα ή έμεσα τον ιατρό ο οποίος θα επιφορτιστεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία και τις διαδικασίες κήρυξης σε αναπηρία ε, που προβλέπει επίσης ε, την μορφή της συμβολιογραφικής πράξης ή την απουσία της συμβολιογραφικής πράξης στην διαδικασία καταγραφής από τις δημόσιες αρχές του πιστοποιητικού αυτού που προβλέπει επίσης σε τους ελέγχους τους οποίους θα πρέπει να, να υφίσταται ο έντολοδόχος που προβλέπει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των ε, επιπτώσεων της συγκεκριμένης πράξης η οποία επικυρώνεται από τις δημόσιες αρχές και καταγράφεται από αυτές και προβλέπει επίσης και την έκδοση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού το οποίο επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του εντολοδόχου του αναπήρου και επιτρέπει την ελεύθερη άσκηση και στο εξωτερικό εκτός χώρας των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το 650 του 2012 ε, στα πλαίσια του πιστοποιητικού για ε, διαχείριση διαδοχής. Νομίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό ο Ευρωπαίος νομοθέτης ε, θα έρθει πιο κοντά στην ανάγκη η οποία υπάρχει και στις επιθυμίες των συμπολιτών μας. Μπορούμε να αυτοκτονήσουμε. Thank you very much, sir. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σαφή αυτά που μας είπατε. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Άνεκε Νεγκόρ, που είναι νομική σύμβουλος ε, σε θέματα διαχείρισης περιουσίας διεθνώς. Είναι μέλος της Commission Levens Testament της Ολλανδίας. Έχετε το λόγο κυρία μου. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, Ευχαριστώ πολύ που, μας, που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω περισσότερα πράγματα για την κατάσταση στην Ολλανδία. Το, είπατε τη λέξη κλειδί. Κομίση Levens Testament. Ε, αυτή δημιουργήθηκε το 2010 από το EPN που είναι ένα τμήμα της Βασιλικής Ένωσης Συμβολογράφων και η ειδική επιτροπή αυτή έπρεπε να επεξεργαστεί πλαίσιο για ένα περίτεχνο μόνιμο πληρεξούσιο που θα λεγόταν Levens Testament. Δηλαδή Levens Testament είναι διαρκές ή μόνιμο πληρεξούσιο. Αυτό το Levens Testament μπορεί να είναι ένα πολύ μακροσχελές έγγραφο αφού καλύπτει ένα σωρό θέματα και δίνει στο πληρεξούσιο το δικαίωμα να χειρίζεται όλα τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα ή χρηματοοικονομικά, δίνει τη δυνατότητα στον πληρεξούσιο να χειρίζεται θέματα ιατρικά, θέματα πρόνοιας, μπορεί να χειρίζεται συγκεκριμένα αιτήματα από τον εντολέα προς τους γιατρούς τους, δικαστές, τον πληρεξούσιο, ε, σχετικά στους ε, γιατρούς, σχετικά με θεραπείες ή μη θεραπείες θέματα ευθανασίας, στους δικαστές όταν πρέπει να αποφασίσουν, για παράδειγμα, όταν ο εντολέας έχει ας πούμε ε, πάθει ένα σοβαρό ατύχημα αλλά ε, έχει μικρά παιδιά και χρειάζεται να οριστεί επίτροπος, τότε καλό θα ήταν ο, ο δικαστής να έχει μια ιδέα ποιον είχε υπόψη του εντολέας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ε, αν ο εντολέας που έδωσε το πληρεξούσιο είναι ο ίδιος επίτροπος μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο είναι ενήλικο αλλά με αναπηρία μπορεί επίσης να φροντίζει έναν γονέα που νοσεί ψυχικά και αν μετά από ατύχημα δεν μπορεί πια να είναι επίτροπος τότε κάποιος θα πρέπει να διοριστεί μετά από εκείνον. Επίσης ο εντολέας ε, μπορεί να ζητήσει ε, από τον ε, πληρεξούσιο να χειριστεί θέματα πώληση του σπιτιού, αν αυτό το επιθυμεί, τι θα γίνει με τα έπιπλα ή με τις συλλογέ ε, γραμματοσύμων. Το Levens Testament δεν τα καλύπτει όλα αυτά τα θέματα, καμιά φορά αναφέρεται μόνο σε ένα θέμα. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ένωση Συμβολογράφων, πάνω από το 80% των Levens Testaments που έγιναν το 2015 κάλυπταν περισσότερα από ένα ζήτημα. Δηλαδή όχι μόνο ιατρικά θέματα ή οικονομικά θέματα μόνο, αλλά συνήθως έπιαναν όλο το πακέτο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχουν ειδικέ διατάξεις στο Ολλανδικό Δίκαιο που αφορούν ειδικά το Levens Testament. Το Levens Testament στηρίζεται στους συνήθεις νομικούς κανόνες των εξουσίων. Το Levens είναι το αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας μιας ομάδας ανθρώπων που ε, κατάλαβαν ότι οι νομικοί και τα ευάλωτα άτομα στην Ολλανδία χρειάζονταν ένα νέου τύπου έγγραφο για να προετοιμαστούν για μια περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο δεν μπορεί πλέον ή δεν είναι σε θέση, δεν επιθυμεί πλέον να φροντίσει τον εαυτό του και τα ε, συμφέροντά του. Το ίδιο ισχύει για το κεντρικό μητρό του Levens Testament, το οποίο ε, άρχισε να λειτουργεί το 2012 και αυτό ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας του ε, EPN, της Ειδικής Επιτροπής ε, και η πρωτοβουλία αυτή ανελήφθη από την Βασιλική Ένωση των Συμβολιογράφων. Η καταχώρηση των, ε, ενός Levens Testament στο κεντρικό μητρό δεν αποτελεί υποχρέωση, γίνεται σε βάση προαιρετική. Μέχρι τώρα το μητρό είναι ανοιχτό σε συμβολιογράφους μόνο, αλλά στο μέλλον θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και δικαστές και γιατροί. Θα μπορούν δηλαδή να ε, ελέγχουν αν κάποιος έχει δώσει οδηγίες για ιατρικές θεραπείες ή ε, το διορισμό των επιτρόπων. Κάθε χρόνο ο αριθμός των ε, εγγραφών αυξάνεται. Το 2015 ήταν περισσότερες καταχωρήσεις κατά 65%. Από το 2012 τώρα οι εγγραφές αυτές, οι καταχωρήσεις έχουν φτάσει τον αριθμό των 135. Η Ολλανδία είναι χώρα διασυνοριακή. Είναι μικρή χώρα. Εγώ μένω στο Άμστερνταμ, πάω προς Ανατολικά με το αυτοκίνητο μια ώρα είμαι στη Γερμανία, ε, προς Νότον μια ώρα είμαι στο Βέλγιο, αλλά και από άλλες απόψεις το διασυνοριακό ζήτημα δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει στην Ολλανδία αφού έχουμε περίπου 17 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων οι 850.000 δεν έχουν εθνικότητα, υπηκότητα Ολλανδική. 3,5 εκατομμύρια κάτοικοι από τη χώρα μου ε, προέρχονται από άλλη χώρα, όχι από την Ολλανδία. Δηλαδή έχουν επαφές, σύνδεση, συνδέσμους με άλλες χώρες, μπορεί να έχουν και ε, περιουσία στην άλλη χώρα. 80.000 νοικοκυριά έχουν δεύτερο σπίτι στο εξωτερικό. Τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια είναι μέσα στην Ευρώπη. Το 2009 41.000 άνθρωποι, 41.000 άνθρωποι έφυγαν από την Ολλανδία για να εγκατασταθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ 64.000 άνθρωποι, αυτά τα πήρα από την, ε, επίσημα στοιχεία, ε, ήρθαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ολλανδία. Ε, κατομμύρια, Ολλανδοί, ναι, ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτά τα νούμερα είναι πολύ σημαντικά για μια μικρή χώρα όπως η Ολλανδία. Κατομμύρια Ολλανδοί πηγαίνουν για διακοπές στο εξωτερικό. Ε, πέρσι αυτό συνέβη 18 εκατομμύρια φορές, δηλαδή ένας πολύ σημαντικός αριθμός Ολλανδών κατοίκων ταξιδεύουν περισσότερο από μια φορά το χρόνο. Ε, το χρόνο. Ε, έχουν περιουσία επίσης πολύ εκτός συνόρων, σπίτια, λογαριασμοί κλπ ε, ή άνθρωποι που κληρονομούν από συγγενείς που δεν ζουν στην Ολλανδία ή άνθρωποι που μένουν σε μια χώρα και εργάζονται σε μια άλλη. Ειδικοί φορολογικοί κανόνες ισχύουν για αυτούς. Ή μπορεί κάποιος να παίρνει τη σύνταξη από άλλη χώρα, όχι από αυτήν που, στην οποία διαμένει ή ε, παίρνουν κάποιο εισόδημα από ασφαλή ζωή που έγινε στο εξωτερικό. Ή κάποιοι πηγαίνουν στο εξωτερικό και παθαίνουν κάποιο σοβαρό ατύχημα και κάποιες ιατρικές αποφάσεις πρέπει να, να ληφθούν στο εξωτερικό. Ε, πρέπει να ανακατευθεί η αστυνομία ξένης χώρας, ε, ε τα δικαστήρια, οι ασφαλιστικές εταιρείες ξένης χώρας ή κάποιος χωρίζει και ο άντρα ε, στη χώρα Α πρέπει να δώσει διατροφή στην πρώην σύζυγο και τα παιδιά στην χώρα Β. Ε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να συμβεί κάποιος άλλος να πρέπει να φροντίσει τα συμφέροντά σας. Όταν δίνετε πληρεξούσια σε κάποιον που εμπιστεύεστε, τότε θέλετε το πρόσωπο αυτό να μπορεί να δράσει, να ενεργήσει για λογαριασμό σας και όταν πρόκειται για θέματα διασυνοριακά. Και ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα από τη δική μου πείρα. Ε, ένα Ολλανδό παντρεύεται μια Αγγλίδα και μένει μαζί τη στην Αγγλία από το 1950. Το ζευγάρι είναι στην ένατη δεκαετία της ζωής τους, ε, δεν, δεν έχει καλή υγεία ο σύζυγος, έχουν ένα παιδί και του έδωσαν μόνιμο, μόνιμο βάσει βάση του Βρετανικού δικαίου. Η κόρη έχει πρόσβαση στο Βρετανικό λογαριασμό τη Τράπεζα του πατέρα, προσπαθεί να έχει πρόσβαση και στον τραπεζικό λογαριασμό τη Ολλανδία. Εκεί πληρώνεται η σύνταξη. Η Ολλανδική Τράπεζα αρνείται να δεχτεί το πληρεξούσιο. Μόνο μετά το θάνατο του πατέρα η χείρα και η κόρα αποκτούν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει να πεθάνει δηλαδή ο πατέρα για να ανοίξει πρόσβαση στο λογαριασμό. Άλλο παράδειγμα. Μια χείρα Ολλανδή ε, μένει μόνη τη στην Ολλανδία, χωρί παιδιά, χωρί άλλου συγγενεί. Είναι 80 ε, και. Κάποιοι καλοί φίλοι, ένα ζευγάρι, ε, την φρόντιζαν κατά τα τελευταία χρόνια. Ε, ε, φροντίζουν τη διαχείριση, το σπίτι της στην Ολλανδία, το εξοχικό της στη Γαλλία. Όταν επιδεινώνεται η υγεία της χείρα και δεν μπορεί να ταξιδεύει στη Γαλλία πλέον, το σπίτι στη Γαλλία πρέπει να πουληθεί. Η χείρα έχει κάνει ένα Levens Testament και όρισε τους φίλους της ως πληροεξούσιους. Το Levens Testament έχει άμεση ισχύ και αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι πληρεξούσιοι μπορούν να πουλήσουν και το σπίτι στην Ολλανδία και το σπίτι στη Γαλλία. Όμως ο Γάλλος συμβολιογράφος δεν θέλει να δεχτεί το Leffens Testament εκτός και αν ε, συνοδεύεται από ένα ιατρικό πιστοποιητικό που λέει ότι δεν είναι ικανή η χείρα για δικαιοπραξία. Άλλο παράδειγμα, ο Ολλανδός με άνω των 80. Έζησε, ε, ε, εργάστηκε στη θάλασσα, ε, δούλεψε για μια ναυτιλιακή Ολλανδική εταιρεία και ζούσε σε μια νοτιοαμερικανική χώρα για πάνω από 30 χρόνια, είναι μόνο, δεν έχει παιδιά, για τα αδέρφια του όλα ζουν στην Ολλανδία πριν από πολλά χρόνια, έδωσε πληρεξούσιο στην αδερφή του που ζει στην Ολλανδία, ούτω ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα συμφέροντά του στην Ολλανδία και να έχει πρόσβαση και στον τραπεζικό λογαριασμό στην Ολλανδία, όπου καταβαλόταν και η σύνταξη. Η αδελφή είναι 75 ετών και θα μπορούσε να πεθάνει ή να νοσήσει ψυχικά. Γι' αυτό ο άνθρωπός μας θέλει να δώσει παρόμοιο πληρεξούσιο ε, στην ανιψιά του, κόρη της αδελφής. Ε, επειδή δεν είναι καλή υγεία, δεν μπορεί να πάει από την Νότια Αμερική στην Ολλανδία. Η αδελφή και η ανιψιά τον επισκέπτονται στην ε, Νότια Αμερική και υπογράφει πληρεξουσιο μπροστά σε έναν ε, ψυμπολιογράφο ε, Νοτιοαμερικανό. Όταν γυρίζει στην Ολλανδία, η Ολλανδική Τράπεζα δεν δέχεται το πληρεξούσιο. Ε, εγώ ε, έχω πολλούς Ολλανδούς ε, πελάτες που έχουν εξοχικά στη Γαλλία ή ζουν στη Γαλλία τους τελευταίους μήνες πάνω από μία φορά. Έπρεπε να αντιμετωπίσω το εξή ζήτημα. Μπορώ να κάνω, μου έλεγαν, ένα Leven Testament το οποίο θα έχει ισχύ και στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Δύσκολο το ερώτημα να απαντηθεί. Όταν το ζευγάρι έχει περιουσία και στις δύο χώρες θα πρέπει να δώσουν δύο πληρεξούσια. Το ένα που θα είναι το Mandate Protection Future στη Γαλλία και ένα Levensestament στην Ολλανδία. Μία κατάσταση παρόμοια με το πρόβλημα που είχαμε πριν από, τον, 17 ε, Αυγούστου του 2015 με τους νόμους ε, κληρονομίας. Δύο διαδοχής, δύο διαφορετικά νομικά συστήματα ε, που εφαρμόζονται στο ίδιο πρόσωπο και στην περιουσία του είναι, γίνεται πιο περίπλοκη ζωή και μέσα από την ψηφιοποίηση της κοινωνίας. Η Ολλανδική κυβέρνηση κινείται προς την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των επαφών με τους πολίτες. Ε, οι νέοι και πιο ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να δουλέψουν με το κομπιούτερ στο τέλος θα είναι ευάλωτοι ενήλικες διότι δεν θα μπορούν να ζητήσουν την ε, βοήθειά τους, τη βοήθεια που λαμβάνουν ή να συμπληρώσουν τη φορολογική δήλωση για να πάρουν αυτά που δικαιούνται, γιατί δεν θα μπορούν να χειρίζονται τους κομπιούτερς. Το Levens Testament δεν λειτουργεί μόνο όταν κάποιος ε, ε, έχει πρόβλημα ε, ψυχικό ή σωματικό. Το Levens Testament όταν ο εντολέας θέλει το λέμε σε να έχει άμεση ισχύ, τότε ο πληρεξούσιος μπορεί να βοηθήσει τον εντολέο όταν η ζωή του γίνει περίπλοκη ε, και για να χειριστεί θέματα εκτός από θέματα υγείας άλλα. Ε, δεν ε, έχει ακόμη επικυρωθεί η συνθήκη της χάγη από την Ολλανδική κυβέρνηση, γιατί είναι μεγάλο το κόστος λειτουργίας κεντρικής αρχής. Νομίζω ότι η αναγνώριση ε, τέτοιων ε, πληρεξουσίων είναι πολύ σημαντικό και η ε, Χάγη 35 θα πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα εφόσον θα ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το δεύτερο θα ήταν να δοθεί να, να, να, να επεκταθεί η Χάγη 35 με μορφή κανονισμού ε, εισάγοντας τη δυνατότητα διεθνούς πιστοποιητικού. Αυτή τη στιγμή η Ολλανδία έχουν 3,5 εκατομμύρια κατοίκους ηλικίας άνω των 65 ετών. Από αυτούς 1,2 εκατομμύρια ε, είναι μόνοι, ε, δεν είναι παντρεμένοι. Κάθε χρόνο οι δικαστές στην Ολλανδία ε, φέρνουν περισσότερες υποθέσεις που θα πρέπει να αποφασίσουν για επιτροπία ή ε, διαχείριση καταπιστεύματος. Μέχρι το τέλος του 2014 η διαχείριση καταπιστεύματος ε, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 240.000 ανθρώπους. Χωρίς έγγραφο, όπως το στις σταμέντε, δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυνατότητες. Αυτά τα πληρεξούσια θα πρέπει να αναγνωριστούν σε διεθνές επίπεδο και γι' αυτό χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το ε, λόγο στον κύριο Φρίμστον, ο οποίος είναι ε, δικηγόρος ε, και ειδικό στο Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα ανέφεραν οι συνάδελφοί μου ήδη, διότι πιστεύω ότι θα ακούσετε διπλούν τα όσα υπόθηκαν, όμως ε, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά το Λονδίνο, το 40% του πληθυσμού γεννήθηκε έξω από το Ηνωμένο Βυσίλειο. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι ζουν σε άλλα κράτη-μέλη και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι να μιλήσω λιγάκι για την ε, Χάγη 35 και για το πώς τη χρησιμοποιούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιες είναι οι διαφορές ε, μεταξύ της Ουαλίας, της κατάστασης στην Ουαλία και τη Χάγη 35, καθώς επίσης και το μίσο που η Χάγη 35 θα μπορούσε να βελτιωθεί. Τα ζητήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε όσον αφορά το ε, διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, είναι ξεκάθαρα. Είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Όσον αφορά όμως την ικανότητα, είναι ζητήματα τα οποία επεκτείνονται σε όλο το εύρος ε, της, ε, του νόμου. Δεν είναι μια συγκεκριμένη νομική κατηγοριοποίηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επεκτείνεται σε ό,τι κάνουμε. Η Χάγη 35 βεβαίως ε, αφορ... Ε, σχετίζεται αποκλειστικά με ζητήματα τα οποία αφορούν τη δικαιοδοσία των εφαρμοστέων νόμα, καθώς επίσης και την αναγνώριση και την εφαρμογή, καθώς επίσης και προστατευτικά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με τον εφαρμοστέο νόμο όσον αφορά σε τομείς ε, της μόνιμης εξουσιοδότησης. Μία από τις βασικές αδυναμίες της Χάγης 35 όμως είναι ότι, ασχολού, ε, ενώ ασχολείται καλά με τα προστατευτικά μέτρα, εκεί λειτουργεί καλά όμως ε, όσον αφορά την εκπροσώπηση και όπως ακούσατε, δεν λειτουργεί τόσο καλά. Πώς λοιπόν χρησιμοποιούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο την hg ε, 35 οι διαφορές μεταξύ ημών ε, και της ε, Χάγης 34 είναι ότι ενώ έχουμε υπογράψει και η Βρετανία έχει επικυρώσει τη Χάγη, το έχει κάνει αυτό μονάχα όσον αφορά τη Σκοτία με αποτέλεσμα ε, η Χάγη 35 να μην, έχει, ε, να μην ισχύει για την Αγγλία. Στην Αγγλία και την Ουαλία εφαρμόζουμε την ίδια νομοθεσία όπως και στις κάτω χώρες, όμως ε, την εφαρμόζουμε σε άτομα τα οποία είναι 18 ετών και όχι 16, εκτός και αν η Χάγη 34 ή οι Βρυξέλλες 2 εφαρμόζονται καλύτερα. Τώρα όσον αφορά τον ορισμό ενηλίκων, η βρυξελλες 2 είναι ξεκάθαρη ότι αυτό εφαρμόζεται μονάχα εάν ένας ε, ε, ενήλικας ε, δεν μπορεί να προστατεύσει τα προσωπικά του συμφέροντα. Όμως εμείς χρησιμοποιούμε τη Χάγη 35 και όσον αφορά τα ζητήματα της εκπροσώπησης όταν ένας ενήλικας λοιπόν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Η τελευταία διαφορά η οποία είναι όμοια με την Αυστρία και την Ολλανδία τις κατοχώρες είναι ότι έχουμε μια αναγνώριση και εφαρμογή τόσο από ε, κράτη τα οποία έχουν επικυρώσει τη Χάγη 35 αλλά και όσον αφορά κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη Χάγη 35 έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε και εφαρμόζουμε προστατευτικά μέτρα από οποιοδήποτε κράτος ε, του πλανήτη το εφαρμόζουμε αυτό παγκοσμίω λοιπόν όμως αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί και ορισμένες δυσκολίες. Είχαμε μια σειρά υποθέσεων στο δικαστήριά μας κατά τη τελευταία δεκαετία ε, που ασχολήθηκαν με τέτοια ζητήματα, δηλαδή το αν η χρήση ε, της Χάγης 35 μεταξύ των συμβαλόμενων και μη συμβαλόμενων κρατών θα πρέπει να είναι διαφορετική και ε, τα δικαστήριά μας κατέληξαν ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται ε, διεθνώς ενώ ταυτόχρονα είχαμε ζητήματα και όσον αφορά ε, την εθνική νομοθεσία είχαμε αρκετούς πολίτες για παράδειγμα από την Ιρλανδία οι οποίοι έρχονται, στην Αγγλία έχοντας στόχο να έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ατροφονομικευτική περίθαλψη η Ιρλανδία λοιπόν τους δίνει επαρκή ε, ε, προστασία και γενικότερα τα δικαστήρια μας έχουν πει ότι δεν θα πρέπει να, να επιβάλλουμε ε, μέτρα εθνικής νομοθεσίας εκτός και αν είναι ακραία. στείλαμε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα στο, στα Ιρλανδικά δικαστήρια ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη τους ερωτήματα όσον αφορά την ε, εκπροσώπωση το αν κάθε άτομο θα πρέπει να εκπροσωπείται και να έχει μια εκπροσώπηση και τα δικαστήριά μας ε, απάντησαν καταφατικά σε αυτό Και για εμάς ε, το άλλο θέμα στο οποίο εφαρμόζουμε τη Χάγη 35 εντελώς διαφορετικά από, το εθνικό, από την εθνική μας νομοθεσία είναι εκεί όπου η εθνική νομοθεσία σχετίζεται με το γεγονός αν κάποιος μπορεί ή όχι να διαχειριστεί τις υποθέσεις του. Ο ορισμός της Χάγης 35 είναι διαφορετικός ε, και εμείς ε, εφαρμόζουμε λοιπόν τον ορισμό της Χάγης 35 άμεσα. Και τέλος, το δύσκολο ερώτημα της συνήθους διανομής, τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την ομοθεσία η συνήθως ε, διαμονή λοιπόν ε, είναι ε, ενιαία σε όλη την Ένωση και έχει οριστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό φυσικά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σχετικά με το που θεωρείται ότι έχει την μόνιμη διαμονή του ένας, ένα άτομο. Το βασικό πρόβλημα το οποίο εγείρεται όμως είναι ε, ε, αφορά ε, την εξουσιοδότηση και ως δικηγόρος θα ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι το 95% των προβλημάτων των πολιτών στον τομέα αυτό δεν σχετίζεται τόσο με την προστασία του ατόμου αλλά σχετίζεται με την πρόσφαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό στην, σε περιουσιακά στοιχεία στην πώληση ενός ακινήτου Εκείνοι που αντιμετωπίζονται τα βασικότερα προβλήματα και συνολικά λοιπόν η Χάγκη 35 εκεί είναι ε, που λειτουργεί πάρα πολύ καλά όσον αφορά τον εφαρμοστέο νόμο, όμως ε, δυσκολεύει στην αποδοχή, στην αποδοχή μιας τέτοιας εξουσιοδότησης με αποτέλεσμα ο πολίτης να μην έχει καμία εναλλακτική από το να δώσει εξουσιοδότηση σε κάθε ε, χώρα όπου έχει εξουσία. Δεν υπάρχει δυνατότητα για την εφαρμογή της ε, εξουσιοδότησης στο πλαίσιο της Χάγης 35 Όσον αφορά λοιπόν την αναφορά αυτή, ε, λέγεται ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ε, εικόνα για αυτό και τώρα δεν φαίνεται αν η εξουσιοδότηση έχει καταγραφεί ε, ή αν έχει συνδεθεί με κάποιο δικαστήριο με αποτέλεσμα να μπορεί να υπάρξει ένα μέτρο προστασίας το οποίο θα σχετίζεται με την εφαρμογή και την προστασία. για πάρα πολλούς εξημών που έχουμε λάβει τέτοια εξουσιοδότηση η ε, ΧΑΚΙ 35 δεν δίνει κάποια λύση. Έχουμε ε, απτές δυσκολίες όσον αφορά την ε, διατήρηση της ε, εγγύησης της εξουσίας αυτού που έδωσε την εξουσιοδότηση. Πολύ συχνά όμως τα πρακτικά προβλήματα προκύπτουν από το άρθρο 14 και ότι ο εφαρμοστέος νόμος δεν ασχολείται με την τοπική εφαρμογή. Η τοπική εφαρμογή της εξουσιοδότησης ορίζεται από το τοπικό νόμο. Ο πελάτης μου δηλαδή που είναι Άγγλος έχει δώσει μια εξουσιοδότηση στην Αγγλία, ζει στη Σκοτία, ο δικηγόρος θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στον γαλλικό τραπεζικό λογαριασμό ο συμβολιογράφος στη Γαλλία λέει ναι, ισχύει η εξουσιοδότηση, όμως ε, υπόκειται ε, στον γαλλικό νόμο με αποτέλεσμα ένας γαλλικός γιατρός θα πρέπει ε, να κάνει εξέταση και να επιβεβαιώσει ότι έχει έλλειψη ικανότητας, τότε στη συνέχεια η εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να καταγραφεί στα γαλλικά δικαστήρια Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έτσι ε, αφαιρούνται πάρα πολλά από τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη της Χάγης 35. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι εμείς που εφαρμόζουμε ε, τη νομοθεσία αυτή ε, θα θέλουμε να δούμε μια νομοθεσία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά είναι, ε, συμφωνούν με την νομοθεσία σχετικά με την κληρονομιά και παρόλο που η Χάγη 35 προέκυψε ύστερα από τη Χάγη 34 σχετικά με την προστασία των παιδιών, ενώ τα ερωτήματα όσον αφορά τα παιδιά είναι ξεκάθαρα, ανήκουν ξεκάθαρα στο οικογενειακό δίκαιο όσον αφορά τη διαχείριση της περιουσίας ένας ε, πολίτη ίσω να μην έχει οικογένεια, ίσω να θέλει να δώσει την εξουσιοδότηση αυτή σε ένα φίλο ή σε ένα δικηγόρο. Με αποτέλεσμα να μην είμαι σίγουρο, εάν όλα αυτά είναι ζητήματα οικογενειακού δικαίου και ίσω λοιπόν θα πρέπει ε, η νομοθεσία να βασιστεί στο άρθρο 81,2. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να δούμε μια, έναν κοινό ορισμό σχετικά με το εύρος της προστασίας, ε, την συνήθεια κατοικία ε, και είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά ε, ώστε να έχουν ε, μια ευρεία εφαρμογή Όπως αναφέρθηκε, η επιλογή της ε, δικαιοδοσίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν έχω το δικαίωμα ε, να ε, δώσω μια εξουσιοδότηση και κατοικώ στην Ισπανία, η οικογένειά μου όμως είναι στην Αγγλία, τότε δεν θα ήθελα να δώσω την εξουσιοδότηση στην Ισπανία, γιατί να μην επιλέξω για παράδειγμα την Αγγλία ως την δικαιοδοσία Ανέφερα επίσης ε, τους περιορισμούς ε, του άρθρου 14. Άλλοι ε, μίλησαν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την αποδοχή και την εφαρμογή των, της εξουσιοδότησης σε όλη την Ευρώπη και επίσης σε περίπτωση που χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΚΝΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για όλα αυτά τα θέματα και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια κινητοποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης ε, σας ευχαριστούμε για την συνεισφορά σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Jean Χριστόφ ε, από τη ΓΑΣ, ο οποίος είναι Γάλλος συμβολιογράφος. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου που συμμετέχω σήμερα στην ακρόαση η οποία οργανώνεται για να μοιραστώ μαζί σας την δική μου μαρτυρία για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου μου στον τομέα της προστασίας των εύθραστων κατηγοριών πολιτών. Θα βασιστώ στην εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει σαν συμβολιογράφο στην Νότια Γαλλία, σε μόνιμη επαφή με ξένους πολίτες πολλών εθνικοτήτων που έρχονται να ζήσουν στην περιοχή μου και μάλιστα να τερματίσουν και τη ζωή τους εκεί. Υπάρχει θέμα διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων, αυτή τη στιγμή ε, ε, καταστούν μη ικανοί να την διαχειριστούν. Η απόκτηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων δεν πρέπει να είναι εμπόδιο σήμερα επί τη βάση της Σύμβασης της Χάγης του 2000 σχετικά με την αναγνώριση αυτών των αδειών των πιστοποιητικών της κυκλοφορίας και της ισχύω τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσω να σας δείξω από κοντά τις αιτίε που με οδήγησαν να εκφραστώ για την προσταχία την διεθνή των ευάλωτων ή έφραστων μάλλον ενηλίκων, πώς έχουν τα πράγματα και πώς η Χάγη 35 παρουσιάζεται σήμερα σαν ευρωπαϊκό μέσο. Αυτή η Διεθνή Σύμβαση εναρμονίζει τους κανόνες σύγκρουσης αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών. Καθορίζει επίσης και την βασική σύνηθη κατοικία του συγκεκριμένου ενήλικα αντί του κριτηρίου της εθνικότητας του διεθνούς ιδιωτικού γαλλικού δικαίου. Ε, επί τη βάση λοιπόν των 5 και 13, άρθρων 5 και 13, οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνε για τη λήψη των αποφάσεων και η εναρμόνιση ακριβώς αυτών των δικαιοδοσιών και των διαδικασιών των νομοθετικών ε, μπορούν να καταστήσουν πιο εύκολη την εφαρμογή των νομικών ρυθμίσεων, ε, των διεθνών ρυθμίσεων, παρά την εφαρμογή ενός άλλου δικαίου όπως του ιδιωτικού εσωτερικού γαλλικού δικαίου, το οποίο ε, επί τη βάση του άρθρου 3 του αστικού κώδικα καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του δικαίου του εδάφους στην Γαλλία. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό μέσω του άρθρου 5.1 μπόρεσα να συμβουλέψω σαν παράδειγμα τα δύο παιδιά των Βρετανικών οικογενειών να καταθέσουν ένα αίτημα ε, στους ε, αρμόδιους περί δικαστές του Μοντομπό. Ο δικαστής επί τη βάση των άρθρων 5.1 και 13 Όρισε την διαδικασία και σύμφωνα με την γαλλική νομοθεσία επέτρεψε την εκκίνηση μιας διαδικασίας κυδαιμονίας. Αλλά η ασθένεια του Αλσχάιμερ κατέστησε ε, ανίκανη την χείρα στην κατοικία της, η χειροτέρευση της υγείας της οδήγησε τα παιδιά της ε, να την ε, παλινοστήσουν στην Μεγάλη Βρετανία σε μια γλώσσα έτσι ώστε να ε, υπάρξει φροντίδα σε μια γλώσσα η οποία θα της ε, ήταν πιο εύκολη. Ε, αν δεν είχε δεχθεί λοιπόν την διαδικασία αυτή, το 5-2 προβλέπει ότι οι αρχές της νέας χώρας στην οποία εγκαθίσταται ο ασθενής είναι αυτές οι οποίες είναι αρμόδιες. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός απέθανε πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τίθεται πάντως το θέμα της εντολής για την κήρυξη ε, του συγκεκριμένου προσώπου ως αδυνάμου. Αυτό το πιστοποιητικό είναι κάτι το οποίο μπορεί να προετοιμάσει ο ενήλικας όσο είναι ακόμα ικανός. Ε, επί τη βάση της προβλεπτικότητας και της πρόληψης. Ε, αυτό καθορίζεται από την νομική ρύθμιση που ισχύει στην χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος και σύμφωνα με το 18 μπορεί να υιοθετήσει μια δικαιοδοσία νομική διαφορετική από την της εθνικότητάς του. Αυτό είναι κάτι που ανταποκρίνεται και στο φαινόμενο το κοινωνικό που ισχύει σήμερα για τη γύρανση του πληθυσμού. Πρέπει βέβαια η εντολή αυτή να κυκλοφορεί και να γίνεται σεβαστή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο γαλλικό θετικό δίκαιο η εντολή μελλοντικής προστασίας, έτσι θα τη λέμε, προέρχεται από τον νόμο του 2007 που τέθηκε σε ισχύ με την ίδια μέρα με τη σύμβαση της Χάγης την 1η Ιανουαρίου του 2009 η γύρανση του πληθυσμού σήμερα είναι βασικό θέμα όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία. Όλοι το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό ενσωματώνοντας ακριβώς αυτό το πιστοποιητικό μη ικανότητα στο νομικό του σύστημα. Στη Γαλλία ο νόμος της 28 Δεκεμβρίου του 2015 επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της εντολής, οι δυσκολίες όμως της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων αυτών εντολών παραμένουν. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τη δυσκολία αυτή. Είναι αλήθεια ότι η γύρανση του πληθυσμού που συνεχίζεται στο μέλλον θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελευθερία διακίνησης των πολιτών. Πώς μπορεί να προβλέψει κανείς ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που είναι θεμέλια του άρθρου 81 της συνθήκης, αν η επιθυμία αυτοδιάθεσης των προσώπων που έχουν καταστεί ευάλωτα αγνοείται, τη στιγμή ακριβώς που το χρειάζονται. Μήπως εδώ φύγουμε την ελευθερία τους. Αυτά τα έφραστα άτομα σήμερα ε, έχουν μια αυτόνομη νομική ζωή και κατέχουν μια περιουσία η οποία πρέπει να καθοδηγηθεί. Η ε, σύμβαση της Χάγης είναι ένα μέσο το οποίο παρέχει λύσεις αλλά έχει και όρια. Το πρώτο όριο είναι το πεδίο εφαρμογής στον χώρο. Ε, όπως είπα πολλές χώρες έχουν υπογράψει τη σύμβαση αλλά εφαρμόζεται μόνο σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φιλανδία, την Εστονία, την Τσεχία και την Ευστρία. Λόγω της έλλειψης του καθολικού χαρακτήρα λοιπόν, μόνες οι βασικές αξίες του κοινού δικαίου παραμένουν σε ισχύ σε όλες τις χώρες. Ας μου επιτρέψετε τώρα να σας δώσω ένα παράδειγμα στα πλαίσια των γαλλοβετανικών σχέσεων και την αδυναμία εφαρμογή σε μια πορτογαλική περίπτωση. Μιλάμε για έναν Πορτογάλο πολίτη που πέθανε στη Γαλλία, άφησε ένα παιδί Πορτογάλο που είναι κάτοικος Γαλλίας, είναι έφραστη κατηγορία και ο δικαστής του Ροντέζ ε, του ζητήθηκε ακριβώς ε, σύμφωνα με τον Πορτογαλικό νόμο, σύμφωνα με το άρθρο του 138 του αστικού κώδικα της Πορτογαλίας. Το άρθρο 38 δεν έχει υπογραφεί και επικυρωθεί, από την Πορτογαλία αλλά με βάση το άρθρο 3 του αστικού γαλλικού κώδικα, το κοινό δίκαιο δηλαδή, και εφαρμόζεται για την προστασία του Πορτογάλου ενήλικα σύμφωνα με τον εθνικό του νόμο. Ο Γάλλος λοιπόν ο δικαστής, ο οποίος κλήθηκε να πάρει την απόφαση, περιμένει με την απόφαση αυτή από τις 12 Φεβρουαρίου του 2015, τότε που κατέθεσα το αίτημα. Πώς λοιπόν σήμερα μπορούμε να βρούμε σύγχρονες λύσεις ικανές να ανταποκριθούν στην διεθνοποίηση του πληθυσμού και πώς μπορεί να μην να εφαρμόζονται αλλά να εφαρμόζεται το άρθρο 3 του αστικού γαλλικού κώδικα που υπάρχει σε ισχύ από το 1804. Αυτό το άρθρο αντιπροσωπεύει πραγματικότητες μακράν της καθημερινότητας και των αναγκών των επαγγελματιών και των πολιτών. Η πολυδιάσπαση των κανόνων, η προσπάθεια για την έβρεση των κανόνων θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια εναρμόνιση του ε, δικαίου στον τομέα των κληρονομιών και για τα θέματα διαζυγίων και ε, διαδοχών κτλ. Έκανα μία θα έλεγα συγκριτική, μάλλον χρησιμοποίησα μία συγκριτική μελέτη εδώ ε, που είχε ζητηθεί από το Κέντρο Συγκριτικού Δικαίου της Λοζάνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέγεται ότι δεν υπάρχει σήμερα επαρκής νομική βάση για μια ενιοποιούσα διαδικασία σε επίπεδο υλικού δικαίου προστασίας των ενηλίκων. Μια παρέμβαση της κοινότητας δικαιολογείται, τεκμηριώνεται αν το καθεστώς προστασίας, διεθνούς προστασίας του ενήλικα δημιουργεί προβλήματα στην διεθνή νομική διαδικασία και την κοινοτική διαδικασία, στην κινητικότητα των προσώπων αυτών και στην κινητικότητα των αγαθών τους. Η παρέμβαση λοιπόν να τεκμηριώνεται και επιβάλλεται εφόσον πρόκειται για το μοναδικό μέσο για τη διασφάλιση της υλικής δραστηριότητας και της νομικής δραστηριότητας των προσώπων αυτών η οποία αλλιώς θα είναι αβέβαιη, θα κοστίζει περισσότερο, θα είναι λιγότερο λειτουργική και ε, θα δημιουργεί προβλήματα στις αρχές της ε, κοινωνίας αυτής, της κοινοτικής αυτής μορφής δημιουργείται μια πολυδιάσπαση νομική, συνοδεύεται από μια έλλειψη ρυθμίσεων διεθνούς προστασίας και από εφαρμογή εντελώς διαφορετικών καθεστώτων που θα πρέπει εφόσον διαπιστωθεί να καταπολεμηθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκπροσώπων της ε, τα δικαιώματα αυτά να επιβεβαιωθούν και ένα ευάλωτος ενήλικς να προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη και με τις ίδιες εγγυήσεις για την ελεύθερη διακίνηση. Ο νόμος του Δεκεμβρίου 2015 λέγεται νόμος σχετικός με την προσαρμογή του δικαίου και της κοινωνίας στη γύρανση. Το πρώτο άρθρο λέει ότι η προσαρμογή της κοινωνίας στη γύρανση είναι βασικός εθνικός στόχος και προτεραιότητα του συνόλου των δημοσίων πολιτικών του κράτους. Τι περιμένουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν πράγματι από το 2009 ο ενήλικας μπορεί να καθορίσει θεσμικά το επίπεδο έλλειψης ικανότητάς του, θα πρέπει από σήμερα να, προσπαθούμε να, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε συγκεκριμένα σημεία σε επίπεδο μορφής και θεωρίας. Καταρχάς, η έλλειψη δημοσιοποίησης της εντολής κήρυξης. Εάν η σύμβαση έχει καινοτομήσει σε σχέση με την εντολή αυτή, δεν προβλέπονται μέσα δημοσιοποίησης έτσι ώστε να γίνει γνωστή και αποδεκτή από άλλες χώρες. Από τις 7 χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση, μόνο η Γαλλία και η Αυστρία έχουν δημιουργήσει ένα ειδικό μητρό δημοσιοποίησης αυτών των εντολών. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα θέσει σε κίνδυνο ακριβώς τις προβλέψεις του ενήλικα και θα καταστήσει εύθραστες ε, τις νομικές λύσεις που επιλέγει. Παράδειγμα, το άρθρο 1259 1259-2 του αστικού γαλλικού κώδικα, ομολογία του νομοθέτη, τι λέει, ο δικαστής μπορεί να διακόψει τις ε, ε, επιπτώσεις ή τις συνέπειες της συγκεκριμένης αυτής εντολής μελλοντικής προστασίας αν η εντολή αυτή τεθεί σε γνώση του αργότερα από την θέση της σε ισχύ. Αυτές ε, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ε, δεν μπορούν να βελτιωθούν αν το καθεστώς δημοσιοποίησης ε, δεν συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός μητρώου. Θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα οι βασικές αρχές. Ήδη από το 2009 το Συμβολιογραφικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο έχει ακριβώς διασυνδέσει με πραγματιστικό τρόπο ε, τα στοιχεία και τα μητρώα διαφόρων κρατών μελών για να υπάρξει βέβαια ένα μη επίσημο και ατελές μητρώο ευρωπαϊκό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάτι το πιο επίσημο. Από πλευράς του Συμβουλίου λοιπόν των Συμβολιογράφων με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπάρχει μια ιστοσελίδα για τα μέτρα προστασίας των ενηλίκων σε 22 χώρες. Αυτές οι εναλλακτικέ λύσεις ενισχύουν την κυκλοφορία της πληροφορίας και της γνώσης αλλά δεν αντικαθιστούν δυστυχώς την ανάγκη του να καταστήσουμε αυτή τη νομική διαδικασία πιο αρμονική στο εσωτερικό της Ένωσης. Απαιτείται λοιπόν μια υπερεθνική θα έλεγα αριθμιστική παρέμβαση για ένα κοινό μητρό σχετικά με την ύπαρξή τους, τη θέση τους σε ισχύ, την τροποποίησή τους, την διακοπή λειτουργία τους ή τη διαγραφή τους. Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη σύστασή του της 9ης Δεκεμβρίου του 2009 λέγει στην αρχή υπαρίθμε 7. Τα κράτη θα πρέπει να ορίσουν με συγκεκριμένο τρόπο τη θέση σε ισχύ της συγκεκριμένης εντολής στην περίπτωση ανικανότητας του εντολέα. Τα κράτη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν τους τρόπους με τους οποίους η συγκεκριμένη αυτή ανικανότητα θα καθορίζεται και θα βεβαιούται. Πρέπει να προτείνουμε επίσης και δύο άλλα πεδία σκέψης. Πρώτον, είναι απαραίτητο και θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους να προβλέψουμε μια δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη Χάγη 35. Δεύτερον, θα μπορούσαμε επίσης ε, να προβλέψουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός μέσου το οποίο θα καλύπτει τις αδυναμίες της σύμβασης αυτής, ιδιαίτερα σε επίπεδο αποδοχής των εντολών αυτών στο εσωτερικό της Ένωσης. Το μέσο αυτό όχι μόνο θα βασίζεται στο υπάρχον και στα μέτρα εθνικής δημοσιοποίησης, αλλά να καλύψει και την απουσία κοινών ορισμών σε επίπεδο κρατών μελών. Το μέσο αυτό θα προσφέρει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην ενίσχυση του σεβασμού της επιθυμίας των ενηλίκων που έχουν καταστεί αδύναμοι επί τη βάση ενός μητρώου κοινοτικού επίπεδου το οποίο θα απαλλάξει αν θέλετε τις διοικητικές και δικαστικές αρχές από την τεράστια προσπάθεια ανείχνευσης ε, της, ε, του ευάλωτου χαρακτήρα το οποίο θα ενισχυθεί στο μέλλον. Θα επανέλθουμε λοιπόν στην εφαρμογή την σωστότερη ε, των ρυθμίσεων της Χάγης 35, γενικεύοντας την εφαρμογή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος όλων, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων ανάμεσά μας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σας για την ομιλία αυτή. Τώρα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Ο κύριος Λορτή μήπως θέλει να μιλήσει. Πριν του δώσω το λόγο πάντως θέλω να καλωσορίσω γιατί το παρέλειψα στην αρχή, την κυρία Μάγια Γκρόφ, που είναι νομική σύμβουλο στη διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Με συγχωρείτε που δεν σας καλωσόρισα στην αρχή και η κυρία Πατρίτσια Ντελούκ από την Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν ίσως θέλει να παρέμβει και να κάνει μια δήλωση για την νομοθετική πρόταση που ελπίζουμε να υποβληθεί εξαρτάται από την Κομισιόν. Ο κύριος Λορτή θέλει να λάβει το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας προσκαλέσατε σε αυτήν την τόσο σημαντική συνεδρίαση θα συμφωνήσουμε με τους εμπειρογνώμοντες που προελάλησαν. Το πιο σημαντικό πρόβλημα σήμερα της Σύμβασης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων είναι ο περιορισμός του χωρικού του πεδίου εφαρμογής, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη κρατική παρέμβαση σε αυτή τη σύμβαση. Πιστεύουμε επίσης ότι μια δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρκετά χρήσιμη βέβαια, θα ήταν καλοδεχούμενη αλλά δεν θα ήταν επαρκής. Θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό μόνο, να πάμε παραπέρα. Να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τη σύμβαση, να βρούμε τους πόρους για να την προωθήσουμε. Μια καλή ιδέα θα ήταν να δημιουργήσουμε σαν παράδειγμα μια διεθνή ε, συνάντηση με ευρωπαϊκές χώρες αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης για την προώθηση της εφαρμογής της σύμβασης, ευαισθητοποίηση των κοινοβουλευτικών στις διάφορες χώρες, ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και όλων επίσης των εμπλεκομένων εταίρων. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη συγκεκριμένη συνεπώς σύμβαση. Υπάρχουν αρκετά, αρκετοί περιορισμοί οι οποίοι ήδη αναφέρθηκαν. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για όρια και περιορισμούς τους οποίους θα χαρακτήριζα θεωρητικούς εν πολλής, διότι ε, με τις λίγες χώρες που έχουν εννέα σήμερα, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα και δεν είμαι βέβαιος ότι τα προβλήματα τα οποία έχουν ε, εντοπιστεί είναι προβλήματα που μπορεί να επιληθούν μόνο σε διακανονιστικό επίπεδο, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και σε πρακτικό επίπεδο οπότε δεν θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, κάτι το οποίο θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο από την έβριση πρακτικών λύσεων. Βρήκα να υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα, στον, ε, ανάμεσα σε δύο ομιλητές για την ελεύθερη κυκλοφορία της συγκεκριμένη εντολής. Αυτή η εντολή αδυναμίας αν θέλετε, η κήρυξη σε αδυναμία καλύτερα, υπάρχουν ε, πολλών ειδών δεν μπορεί να εναρμονιστούν πλήρως, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν εντελώς διαφορετικές νομοθετικές ε, παραδόσεις. Υπάρχουν εντολές κηρύξεις οι οποίες δεν πρέπει να επικυρωθούν από αρμόδια αρχή. Αυτές εντάσσονται στο άρθρο 15 της Σύμβασης και κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες όπως και κάθε άλλη μορφή εντολής ή κάθε άλλη σύμβαση διεθνούς δικαίου. Ε, η κυρία Ντεμασκελή είπε ότι η εντολή αυτή δεν εντάσσεται στο κεφάλαιο 4 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση και εφαρμογή. Ενώ ο κύριος Φερσμιντ είπε ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κεφάλαιο 4. Πράγματι κάποιες ε, τέτοιου είδους εντολές όπως αυτές που γνωρίζουμε στην Ιαπωνία ή στον Καναδά ε, πράγματι υπόκεινται στην επικύρωση από αρμόδια αρχή, δικαστήριο, ή ε, μια δημόσια υπηρεσία όπως ο δημόσιος ε, αρρωγέας ή διαμεσολαβητής, ένα είδος διαμεσολαβητή. Η απόφαση λοιπόν της αρμόδιας αρχής είναι ένα μέσο προστασίας που εντάσσεται στα πλαίσια του άρθρου 3 ε, που μπορεί λοιπόν να γίνει αντικείμενο αμοιβαίας εφαρμογής στα πλαίσια του 22. Δεν νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό αναφέρθηκε από τον κύριο Νταμασέλη. Σχετικά τώρα με την ελεύθερη κυκλοφορία σημειώθηκε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βρούμε κάποιους μηχανισμούς για τη δημοσιοποίηση αυτών των εντολών ε, κήρυξης ή να καθίστανται δημόσιες ε, έστω και μέσω ενός μητρώου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει ένας διεθνής κανόνας για να γίνει κάτι τέτοιο. Στην Γαλλία σαν παράδειγμα υπάρχει ένα τέτοιο μητρό με βάση τον εθνικό νόμο. Και αν πράγματι πρέπει να αμφισβητήσουμε εμείς την ύπαρξη μιας τέτοιας εντολής, μπορούμε να αναζητήσουμε το γαλλικό μητρό. Μιας και όλες οι χώρες κάποια στιγμή θα πρέπει να προβλέψουν τέτοιου είδους μητρώα, στον σύγχρονο κόσμο της πληροφορικής θα ήταν πάρα πολύ απλό να συνδέσουμε όλα τα δίκτυα Μητρώα και να οδηγηθούμε σε μια ενιαία πλατφόρμα χωρίς να έχουμε νομοθετικές ανάγκες. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση, την εφαρμογή της στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης και έτσι θα επιληθούν κάποια από τα προβλήματα όπως είπε η Ολλανδή εκπρόσωπος που είπε ότι έχουμε ανάγκη από διαφορετικές εντολές σε διαφορετικές χώρες. Το ίδιο ισχύει για την Ολλανδία γιατί δυστυχώς η Ολλανδία δεν συμμετέχει στην σύμβαση του 2000. Αν ήταν στη σύμβαση του 2000 το πρόβλημα αυτό δεν θα υπήρχε. Σχετικά με το πιστοποιητικό αυτό το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38. Μα είπατε ότι δεν υπάρχει ειδική διαδικασία, ότι δεν προβλέπετε τίποτα εδώ έτσι ώστε η αμφισβήτηση ε, να ε, κοινοποιείται. Είναι απλός ο λόγος. Όταν ένα κράτος προβλέπει την έκδοση ενός τέτοιου πιστοποιητικού, αυτό γίνεται επί τη βάση του νόμου της χώρας και επί τη βάση του νόμου μπορεί να αμφισβητηθεί το πιστοποιητικό αυτό ή εντολή αυτή. Αυτά είναι θέματα απλά τα οποία δεν απαιτούν περαιτέρω νομοθετικές υπερεθνικές ρυθμίσεις. Στα πλαίσια της διάσκεψης της, της σύμβασης της Χάγης ε, μπορήσαμε λοιπόν να λύσουμε κάποια τέτοια θέματα χωρίς περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήσαμε διάφορους οργανισμούς επαγγελματικούς και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την δυνατότητα τα δίκτυα των συμβολιογράφων στην Ευρώπη από κοινού με οργανισμούς όπως το ΣΤΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο να βρουν λύσεις έτσι ώστε να μπορούμε να διαβουλευόμεθα κάποια μητρά, όχι διακυβερνητικά, αλλά επαγγελματικών οργανώσεων όπως των συμβολεογράφων, για να μπορούμε να εξετάζουμε τις εντολές αυτές και τα πιστοποιητικά. Ε, ταυτόχρονα μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να υπάρξει ένα πρότυπο διακήρυξης σε αδυναμία που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 25 χρόνια υπάρχουν κάποια κοινά πρότυπα και όταν βλέπουμε τα κοινά αυτά πρότυπα δεν τίθενται, δεν υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με τη μορφή τους και αναγνωρίζουμε άμεσα τα συγκεκριμένα έγγραφα. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια αναφορά με μια ιστοσελίδα που θα μας επιτρέπει ε, να, ε, να εξετάζουμε τη συγκεκριμένη εντολή. Δεν απαιτείται νομική ρύθμιση εδώ. Όλα αυτά τα πρότυπα έγγραφα μπορούν να αναπτυχθούν και εφόσον υιοθετηθούν από τα κράτη να κυκλοφορούν ελεύθερα. Μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις ε, ε, είναι στο επίπεδο των πιστοτικών ιδρυμάτων και της ιδιοκτησίας. Και εδώ είτε αναπτύξουμε νέους κανόνες, είτε παραμείνουμε στην διάσκεψη, στη σύμβαση του 2000, νομίζω ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις τράπεζες και να τις ευαισθητοποιήσουμε. Οι τράπεζες όταν έχουν μπροστά τους μια τέτοια εντολή κήρυξη σε αδυναμία, είτε εφαρμοστεί είτε όχι, έχει πάντα κάποιες απορίες και δισταγμούς. Και θα ήταν πάντα χρήσιμο να ευαισθητοποιήσουμε τις τράπεζες για τη χρήση αυτών των μέσων. Κλείνοντας και γνωρίζοντας ε, τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους ε, τα κράτη-μέλη της Σύμβασης της Χάγης, μιας και τα τελευταία δέκα χρόνια συγκεντρώνονται ε, στην ε, εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών, βλέπουμε ότι κάποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για την εργασία μας στον τομέα της Σύμβασης 2000 και το Μονακό συμμετέχει εδώ και δύο εβδομάδες και ξέρουμε ότι και η Πορτογαλία θα πάρει μέρος όπως και η Ιρλανδία κατά τη διάρκεια του 2016. Μας ενημέρωσαν επίσης ότι και η Σουηδία θα πρέπει να γίνει μέλος το 2017. Δεν έχουμε κανένα λόγο λοιπόν να πιστεύουμε ότι η ηγετική θέση των κρατών αυτών δεν θα ακολουθηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας και έχουμε περιορισμένους πόρους λοιπόν θα ήθελα να συζητήσω να είστε επιφυλακτικοί για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα να πιέσουμε τα κράτη να εργαστούν για την εφαρμογή της σύμβασης. Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Είμαστε διατεθειμένοι να δημιουργήσουμε μια διεθνή επιτροπή, αν θέλετε, μια διεθνή συνάντηση τακτική για τα θέματα της σύμβασης, οπότε όλες οι χώρες που θα συμμετέχουν θα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και θα ζητούν και από τα υπόλοιπα κράτη να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Στα λίγα λεπτά που μας μένουν θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη πρώτα, αν έχουν απευθύνουν ερωτήσεις στους διακεκριμένους ομιλητές και μετά να ρωτήσω και την Κομισιόν αν η κυρία Αντελούκα θέλει να παρέμβει. Και μετά η κυρία Μπερζερόν θα κάνει τις καταληκτικές, θα κάνει το κλείσιμο. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας. Κάποιοι ζητούν να δημιουργηθεί ένα νέο μέσο. Κάποιοι υπερασπίζονται τη σύμβαση της Χάγης. Υπάρχει και ενδιάμεση θέση, και σύμβαση και ενδιάμεσο μέσο. Πριν να καταλήξουμε κάπου, θα ήθελα να μου εξηγήσετε ίσως ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο από το 2000 τα κράτη-μέλη δεν έχουν επικυρώσει Επτά μόνο του έχουν κάνει αυτό, δύο θα το κάνουν σύντομα. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους μέχρι τώρα δεν έχει επικυρωθεί σύμβαση. Έχετε κάποιες ιδέες. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητεί άλλος βουλευτής το λόγο. Ποιος θα απαντήσει. Εσείς. μπορώ να απαντήσω επί τη βάση των γνώσεων που έχουμε για τα κράτη-μέλη. Οι πόροι που είναι στη διάθεση των κρατών μελών στα πλαίσια του διεθνούς ιδιωτικού είναι περιορισμένοι. Ήδη από το 2000, από τότε που τέθηκε σε ισχύ δηλαδή η συνθήκη του Άμστερνταμ, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες εδώ στις Βρυξέλλες στον τομέα του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και αυτό έχει, απαιτήσει, έχει απαιτήσει πολλούς πόρους από πλευράς των κρατών μελών. Ε, έχουμε το παράδειγμα της Ιταλίας σαν παράδειγμα, μόλις επικύρωσαν τη σύμβαση του, του, την προηγούμενη σύμβαση το προηγούμενο καλοκαίρι και από τότε ξεκίνησαν να εξετάζουν τη σύμβαση του 2000. Αναφέρθηκα στη σύμβαση του 1996. Ε, υπάρχουν εννέα χώρες που συμμετέχουν στη σύμβαση του 2000. Η τελευταία που μπήκε είναι το 13 η Αυστρία και το Μονακό πριν δύο εβδομάδες. Βλέπουμε τώρα ότι οι επόμενες φάσεις, τα επόμενα στάδια ε, είναι στάδια τα οποία αφορούν χώρες που έχουν θέσει σε ισχύ τη σύμβαση του 1996 πρόσφατα. Ο βασικός λόγος που εξηγεί λοιπόν την καθυστέρηση είναι αυτός. Άκουσα να λένε ανεπίσημα χείλη ότι ορισμένες χώρες, και το ακούσαμε επίσης και από την Ολλανδή εκπρόσωπο, είναι διστακτικές γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εσωτερική ε, διευθυντική αρχή και απαιτούνται πόροι. Οι πόροι είναι περιορισμένοι. Είτε νομοθετούμε εδώ στις Βρυξέλλες είτε στη Χάγη, οι πόροι που απαιτούνται είναι ίδιοι. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Άκουσα επίσης να λέγεται ότι κάποιες χώρες είναι δικα... Ε, διστακτικές γιατί η εφαρμογή της σύμβασης του 96 κόστισε περισσότερο από ό,τι είχαν προβλέψει. Έχουμε χώρες που εφάρμοσαν όμως τη σύμβαση του 2000 και τα θέματα τα οποία χρειάστηκε να καλυφθούν στα πλαίσια της σύμβασης του 2000 είναι πολύ λιγότερα από την αντίστοιχη σύμβαση του 1996 και είναι επίσης θέματα τα οποία δεν έχουν την ίδια ανάγκη δημοσιοποίησης και ανταπόκρισης στα μέσα ενημέρωσης κτλ. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι ε, και τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που γνωρίζουμε η Επιτροπή. Χωρίς... Δεν ακούγεται. Sorry, it seems that... Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Κάποιο πρόβλημα έχει το αυτό το μικρόφωνο. Αυτό το μικρόφωνο έχει πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν ακούγεστε. Ε, χρησιμοποιήστε άλλο μικρόφωνο, παρακαλώ. Αυτό είναι καλό. Ευχαριστώ. Κι άλλες φορές έχω πει στην Νομική Επιτροπή ότι η Κομισιόν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν στην ε, σύμβαση της Χάγης από, ήδη από το 2008 και πολλές φορές κάναμε διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα αστικά θέματα και τα γενικά ζητήματα. Συζητήσαμε δηλαδή τους λόγους μη επικύρωσης και μιλήσαμε και για την πρώτη εμπειρία από την εφαρμογή Αυτά μας τα είπαν βεβαίως τα κράτη που επικύρωσαν τη σύμβαση. Κάναμε λοιπόν αυτή την έρευνα το 10, το 14 και το 15 και σχεδιάζουμε να την επαναλάβουμε φέτος. Η απάντηση των κρατών μελών είναι παρόμοια με αυτή που ανέφερε και ο κύριος Λορτή τώρα μόλις. Πρώτον είναι το θέμα του κόστους διότι φοβούνται ότι η θέσπιση και κεντρικής αρχής συνεπάγεται κόστος για τα κράτη-μέλη. Δεύτερο είναι ο μικρός αριθμός των υποθέσεων. Αφού τα κράτη-μέλη που ήδη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση ανέφεραν στην Κομισιόν πολύ λίγες τέτοιες υποθέσεις και αιτήσεις που ε, δόθηκαν ή λήφθησαν από το άλλο συμβαλόμενο μέρος, μάλλον γιατί είναι λίγα ακόμα τα συμβαλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Χάγης. Και για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν, σχεδιάζουμε φέτος να μεταφράσουμε το επεξηγηματικό μνημόνιο στη, τη Σύμβαση της Χάγης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όχι μόνο αγγλικά, γαλλικά που είναι ε, οι επίσημες γλώσσες της διάσκεψης της Χάγης και σκεπτόμαστε να κάνουμε και κάποιες άλλες δραστηριότητες προώθηση της ε, ε, κύρωσης της σύμβασης. Για μας η σύμβαση είναι καλή, μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα είναι, θα ήταν πρόωρο τώρα να σκεφτούμε να, ε, την ενδεχόμενη ανάληψη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν αυτά να παρουσιαστούν ως θέματα οικογενειακά και γι' αυτό θα προϋποτίθεται ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και τώρα η εισηγήτρια η κυρία Μπερζερόν θα κάνει ένα σύντομο κλείσιμο ή δυνατόν. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι έχουμε την κατάσταση των πραγμάτων πλέον, τη σημερινή κατάσταση. Γυράσκει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, Η Ολλανδή εκπρόσωπος μας έδειξε την σημασία του φαινομένου. Αντίθετα από αυτά που ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις προσώπων διασυνοριακών οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και πέφτουν σε ζώνες μη εφαρμογή του δικαίου. Έχουμε ενήλικες οι οποίοι είναι και ευπαθείς, δηλαδή έχουν κάποια ανεπάρκεια προσωπική και οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά του σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και βρίσκονται και σε διαμεθοριακές ή ε, διασυνοριακές καταστάσεις, δηλαδή ε, προέρχονται από μια χώρα της Ένωσης αλλά κατοικούν τακτικά σε μια άλλη. Όλοι αυτοί οι πολίτες αξίζουν ε, του σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, της βούλησής τους. <coughs> Πρέπει να διασώσουμε τα συμφέροντά τους και η βασική ιδέα είναι οι εθνικές ρυθμίσεις να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο μέτρο ειδικών για τους ευπαθείς και ευάλωτους ενήλικες που δεν εφαρμόζονται δυστυχώς παρά μόνο σε αυτούς οι οποίοι ε, μένουν σε μια χώρα είτε είναι πολίτες της χώρας είτε είναι ξένοι οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ σε σχέση με, ε, τη μελλοντική προστασία ε, και αν αλλάξει η χώρα το προστατευόμενο πρόσωπο όπως μας είπε ο Γάλλος συμβολιογράφος ένας Άγγλος ο οποίος ε, γίνεται προκεχωρημένης ηλικίας και πρέπει να επανέλθει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια άλλη χώρα εκτός Γαλλίας και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει, δεν τον ακολουθεί αν θέλετε ο φάκελός του μέσω του οποίου έχει ε, κηρυχθεί ε, στην ε, ευπαθή κατηγορία. Η σύμβαση της Χάγης του 2000 λοιπόν είναι ένα πολύ ικανοποιητικό μέσο, δεν το έχουν επικυρώσει πολλές χώρες. Λόγω του μικρού, του χαμηλού επίπεδου των επικυρώσεων εφαρμόζεται με περιορισμένο τρόπο ε, χωρικά. Όσο και πραγματιστική και ενδιαφέρουσα να είναι η Συμφωνία της Χάγης, η Σύμβαση της Χάγης, δεν υπάρχει αναγκαστικό μέσο εφαρμογής ακόμα και στις χώρες που την έχουν υπογράψει. Ε, θα μπορούσε να υπάρξει μια επικύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος των κρατών μέλων, αλλά κάτι τέτοιο είναι νομικά εφικτό ένας ευρωπαϊκός κανονισμός ενσωματώνοντας τη σύμβαση της Χάγης θα καταστήσει τη σύμβαση κοινοτικό δίκαιο άμεσα εφαρμόσιμη σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ μια οδηγία θα ήταν λιγότερο υποχρεωτική. Το ευρωπαϊκό δίκαιο θα ήταν επίσης πιο ευέλικτο, θα μπορούσαν μέσω της νομοθετικής διαδικασίας να υπάρχουν αλλαγές χωρίς να αλλάζουν οι διεθνείς συμφωνίες οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν αλλαγές. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις που είναι απαραίτητος, όπως ο ρόλος και ο ορισμός του κηδεμόνα, της εκπροσώπησης, των διαδικασιών για την έκδοση μελλοντικής προστασίας, εντολών μελλοντικής προστασίας και της εγγραφής σε ειδικά μητρώα. Γιατί να μην έχουμε ευρωπαϊκό δίκαιο εδώ μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια διεθνή σύμβαση. Τελειώνοντας, τίθεται ένα ερώτημα. Ένα, μια δικαστική υπηρεσία θα μπορούσε να είναι αρμόδια σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πρέπει να έρθει ακόμα πιο κοντά στους πολίτες. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και οι επαγγελματίες του δικαίου όπως οι συμβολιογράφοι οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά ασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια με την τύχη των ευπαθών προσώπων. Η έκθεση του Λόπες ή του του 2008 δεν έχει εφαρμοστεί. Οι ευπαθείς όμως εξακολουθούν να ζουν με δυσκολίες, ο αριθμός τους αυξάνεται και αυτοί που ζουν ανάμεσα σε δύο χώρες επίσης αυξάνονται. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια εσωτερική αγορά, είναι επίσης ένα κράτος δικαίου. Είναι απαραίτητο το δίκαιο να γίνεται σεβαστό, η αξιοπρέπεια των προσώπων των ευπαθών ιδιαίτερα πολιτών να γίνεται και αυτή σεβαστή. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους Καταλαβαίνω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ όλους εδώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Okay. Uh, Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα στο πέμπτο σημείο της σημερινής διάταξης, το οποίο αφορά την ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Ελένε Βέντλαντ, ε, που είναι αντιπρόσωπος ε, ε, σχετικά του γραφείου του ΙΠΑ του Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το έργο λογοδοσίας και επανόρθωσης. Έχουμε μαζί μας νομίζω και την κυρία Τζένιφερ Σάρκ η οποία είναι ε, τεχνική ε, νομική ειδικό ε, πάνω στο ζήτημα. Κυρία μου, κυρίες μου, ποια θα ήθελε να πάρει πρώτο, πρώτη το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα περιμένω λιγάκι για να φύγει ο κόσμος. All right. Ωραία λοιπόν και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Επιτροπή που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να ε, παρουσιάσουμε ε, το έργο λογοδοσίας και επανόρθωσης ε, σε αυτή την πολύ σημαντική επιτροπή. Το όνομα μου είναι Λένε Wetland Είμαι ε, εκπρόσωπος ε, του ε, γραφείου του ΥΠΑ του Αρμοστή Ηνωμένων Εθνών και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μαζί μου είναι η κυρία Δόκτωρ Τζένιφερ Τζέρκ η οποία είναι σύμβουλός μας σχετικά με την εξέλιξη του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτό το απόγευμα λοιπόν θα σας δώσουμε μια σύντομη εικόνα του ε, ε, προγράμματος καθώς επίσης ε, και ένα σχέδιο της διαδικασίας και του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε τώρα καθώς επίσης και τα αποτελέσματα τα οποία θα παρουσιαστούν φέτος τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η Τζένιφερ θα σας δείξει στη συνέχεια μια παρουσίαση που θα είναι πιο αναλυτική σχετικά με τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και καλωσορίζουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας ε, σχετικά με την οδηγία αυτή. Ε, πολύ σύντομα το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο του να ενισχύσει την πρόσβαση στις ε, επανορθώσεις καθώς επίσης και την ε, λογοδοσία, ιδιαίτερα σε θύματα τα οποία αφορούν κυρίως υποθέσεις των πιο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, έχει ως στόχο να υπάρξει μια πιο εις εφαρμογή των αρχών του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία υποστηρίχθηκαν μάλιστα και το 2011 από την Ολομέλεια του ΟΗΕ. Και όποιος δεν γνωρίζει τις ε, κατευθυντήριες αρχές, αυτές αποτελούνται από τρεις πυλώνες, αρχές, από τρεις πυλώνες αρχών και ο τρίτος πυλώνας αφορά ε, τις επανορθώσεις ε, και συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερως τα κράτη, τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να υπάρχει λογοδοσία αλλά και επανόρθωση. Το ε, πρόγραμμα λογοδοσίας ε, και επανόρθωσης ε, επικεντρώνεται κυρίως σε νομικές επανορθώσεις παρόλο που υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επανορθώσεων όπως είναι οι μη δικαστικές επανορθώσεις. Όμως επειδή η, επειδή η πρόσβαση στη δικαστική επανόρθωση σύμφωνα με τις ε, αρχές του ΟΗΕ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επανορθώσεων. Νομίζουμε, ε, θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε ένα ένα πρόγραμμα, ένα έργο και στη συνέχεια να προωθήσουμε την εφαρμογή αυτών των αρχών ενώ ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε στις, ανησυχίες, στις ανησυχίες που έχουν διάφορα θύματα σχετικά με τα ε, νομοθετικά εμπόδια τα οποία αντιμετωπίσουν για την πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Όμως ε, η επικέντρωση αυτή ε, στις επανορθώσεις δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας άλλες επανορθώσεις, αλλά αφορά κυρίως τον περιορισμό της, του μεγάλου εύρους που έχει το πρόγραμμα αυτό το έργο λογοδοσίας και επανόρθωσης ε, κεντρώνεται σε καλές εναλλακτικέ και πρακτικές για τα κράτη, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στις επανορθώσεις, καθώς επίσης η διαδικασία την οποία αναπτύξαμε από την αρχή του προγράμματος ήταν η συλλογή αποδείξεων ούτω ώστε οι κατευθυντήριες που θα δώσουμε στη συνέχεια να βασιστούν ε, σε απτά ε, στοιχεία σχετικά με το τι λειτουργεί και τι όχι. Ε, καν, είχαμε μια διαδικασία όπου συμμετείχαν διάφοροι παράγοντες με αποτέλεσμα να λάβουμε προτάσεις από κυβερνήσεις, από ε, από επιχειρήσεις, από ειδικού, ε, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι κατευθυντήριες ε, οι οποίες θα δοθούν προς τα κράτη-μέλη να αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων. Οι κατευθυντήριες αυτές θα στοχεύουν σε δράσεις, δεν αφορά απλά ε, το να έχουμε μια καινούργια αναφορά πάνω στο ζήτημα, αλλά ο βασικός στόχος είναι να έχουμε ε, κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες ε, τα κράτη αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν με έναν πρακτικό τρόπο. Το έργο αυτό λοιπόν δεν θα ανταγωνιστεί αλλά έρχεται να προσθέσει σε άλλες πρωτοβουλίες του ΟΗΕ ε, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι για παράδειγμα η ομάδα εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ομάδα εργασίας η οποία ορίστηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μια διακυβερνητική διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2015 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει την εντολή να δημιουργήσει ένα δεσμευτικό ε, πλαίσιο ενώ έχουμε ε, και μια πιο ε, διευρυμένη ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ όπου το έργο λογοδοσίας ε, και επανόρθωσης θα μπορέσει να έρθει να προσθέσει σε όλα αυτά. Το έργο λοιπόν ξεκίνησε το Μάιο του 2013, οπότε και ξεκινήσαμε εξετάζοντας ε, μια ερευνητική διαδικασία σχετικά ποια είναι τα πρακτικά και νομοθετικά εμπόδια για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία η οποία θα σχεδιάσουμε θα ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα σε αντίθεση με αυτά τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά. ένα χρόνο ε, μετά την έναρξη του προγράμματος, ε, το οποίο μάλιστα ε, ξεκίνησε ύστερα από εντολή του γραφείου του ΥΠΑΣ Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνώρισαν το, το έργο αυτό και μας έδωσαν την εντολή να συνεχίσουμε και αυτό λοιπόν θα κάνουμε σε μια τελική αναφορά μέσα στο 2016. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαδικασίας στην οποία βρισκόμαστε τώρα την τελευταία φάση δηλαδή πριν από την αναφορά ε, έχουμε θέση ε, σε διαβούλευση το ζήτημα αυτό ε, ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι θα συζητηθούν στην Επιτροπή και επιζητούμε σχόλια καθώς καθώς σχεδιάζουμε αυτή την τελική αναφορά. Κάποια, αναφορέ ε, κάποιες αναφορές όσον αφορά τη διαδικασία είχαμε διαβουλεύσεις, είχαμε συναντήσεις με ειδικού, είχαμε ε, διαβουλεύσεις όμως ε, πάνω από όλα αυτά υπήρχε μια διαδικασία που ε, περιελάμβανε τη συλλογή ε, δεδομένων παγκοσμίως που έγινε το 2015 και είχαμε μια παγκόσμια έρευνα προσπαθώντας να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες και τις δυσκολίες των εθνικών νομικών συστημάτων ε, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε τι όντως συμβαίνει στα διάφορα μέρη του πλανήτη, να μάθουμε και να ξέρουμε τι λειτουργεί και τι όχι, να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε που είναι τα ε, κενά. Και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είχαμε ε, αναλυτικές πληροφορίες από 130 ε, είχαμε 130 απαντήσεις ε, και έχουμε αναλυτικές ε, λεπτομέρειες από 60 διαφορετικές δικαιοδοσίες σε όλο τον πλανήτη και στην πίτα που βλέπετε είναι λίγο δύσκολο να τη διαβάσετε από εδώ κάτω που βρισκόμαστε όμως αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερως είναι οι ανταποκρίσεις που λάβαμε προέρχονταν από, ε, είχαν μια καλή ένα καλό γεωγραφικό έβρος οπότε μπορούμε να έχουμε την σιγουριά ότι οι κατευθυντήριες τις οποίες θα δώσουμε θα βασίζονται σε δεδομένα που δεν προέρχονται από ένα μικρό πλαίσιο δικαιοδοσιών ε, και νομικών παραδόσεων, αλλά θα αντικατοπτρίζει μια παγκόσμια κατάσταση ενώ είχαμε μια ποικιλομορφία ενδιαφερομένων οι οποίοι συνεισέφεραν στη διαδικασία. Δεν λάβαμε λοιπόν πληροφορίε ε, και δεδομένα μονάχα από μια ομάδα δεν ενδιαφερομένων, αλλά είχαμε ανταποκρίσει από ε, όλες, όλους τους ε, σχετικούς ενδιαφερόμενους. Το πλαίσιο, λοιπόν, πριν η Τζένιφερ μπει σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω άμα είχατε την ευκαιρία να επεξεργαστείτε ε, το έγγραφο το οποίο ε, κυκλοφόρησε, όμως ε, το φορμάτ το οποίο επιλέξαμε ούτως ώστε να είναι λειτουργικό και να μπορέσουν να το υιοθετήσουν εύκολα τα κράτη βασίζεται στα έξι θέματα τα οποία καλύπτουμε. Έτσι δημιουργήσαμε τους στόχους της πολιτικής, της, τους πολιτικούς στόχους, ε, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε δηλαδή όσον αφορά τη λογοδοσία και τις επανορθώσεις, ποιες είναι οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ε, στα εθνικά νομοθετικά συστήματα ούτως ώστε να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητα για τους πολίτες. Θέσαμε λοιπόν τους ε, στόχους, τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε στα έξι διαφορετικά προγράμματα τα οποία έχουμε Κάθε ε, στόχος λοιπόν κατευθύνει τα κράτη για την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, και έχουμε στοιχεία καλής πρακτικής ε, των κρατών στις, στους διάφορους στόχους. Είναι πιο εύκολο να το καταλάβετε άμα το διαβάσετε. Ελπίζω τουλάχιστον γιατί είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω όμως ε, η ιδέα είναι το να δώσουμε ποιος είναι ο στόχος και στη συνέχεια ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να σας κατευθύνουν ώστε να πετύχετε αυτό το στόχο. Και τέλος, με βάση τις αποδείξεις, τις, ε, τα δεδομένα και τις συζητήσεις που είχαμε θα δώσουμε όπου αυτό μπορούμε να το κάνουμε ε, παραδείγματα και περαιτέρω επεξηγήσεις για να μπορέσουμε να δείξουμε το πώς οι καλές πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή. Αυτό θα είναι ανώνυμο βέβαια, δεν θα αναφερόμαστε σε μεμονωμένα κράτη, δεν θα λέμε ότι σε αυτή τη χώρα έκαναν αυτό. Απλά ε, θα δίνουμε αυτά τα παραδείγματα για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε περαιτέρω αλλά και να δείξουμε το πώς αυτές οι κατευθυντήριες μπορούν να εφαρμοστούν τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις κατευθυντήριες και να τις εφαρμόσουν είτε συνολικά είτε μεμονωμένα. Σε ε, ένα λεπτάκι θα ακούσετε ότι υπάρχουν συνολικά έξι σημεία τα οποία καλύπτονται και φυσικά το ένα συμπληρώνει το άλλο. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα θα προέλθουν από, ε, το, ε, λαμβάνοντας δράση σε όλους τους έξι τομείς όμως ένα κράτος μέλος ίσως να επιλέξει να επικεντρωθεί σε ένα μονάχα σημείο λαμβάνοντας ε, κατευθυντήριες από αυτήν, ε, αυτή την ε, επίδειξη την οποία θα έχουμε κάνει. Η εφαρμογή βέβαια μπορεί να γίνει μέσω εθνικών διαδικασιών, αυτό είναι ο πρόσθετος στόχος Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ήδη εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης ε, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων, ενώ υπάρχουν ε, μεταξύ αυτών ε, και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε η Κομισιόν το 2011, τέσσερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτό, όμως υπάρχουν διαδικασίες και σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να εφαρμοστούν για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της εφαρμογής. Αυτό στο οποίο λοιπόν στοχεύουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν μια κατευθυντήριο σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τη λογοδοσία ε, και την επανόρθωση. Αυτό δεν αφορά μονάχα τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και άλλους τομείς και θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα, ότι, ε, έχει έρθει ώρα που νιώθουμε ότι με το πρόγραμμα αυτό ε, θα μπορέσουμε πράγματι να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιτύχουν το συγκεκριμένο στόχο. Έχουμε λοιπόν τη διαβούλευση η οποία συνεχίζεται μέχρι την 1η Απριλίου. Καλούμε ε, όλους ε, τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ε, στη συνέχεια θα υπάρχει ένα ε, έγγραφο, υπάρχει ένα έγγραφο μαζί ε, το οποίο δίνει καλύτερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά και πολύπλοκα ζητήματα τα οποία καλύπτονται στο πρόγραμμα αυτό και θα εξετάσουμε όλα τα δεδομένα τα οποία θα λάβουμε και στη συνέχεια θα κάνουμε τροποποιήσεις των προτάσεων και θα το παρουσιάσουμε εν τέλει στο, ε, στο Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζέκερ η οποία θα αναφερθεί ε, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λένη. Εδώ βλέπετε τις έξι συνιστώσεις που έχουν εξεταστεί στα πλαίσια αυτού του έργου θα τις δούμε μία-μία. Η πρώτη είναι ε, δοκιμές σε εθνικό επίπεδο για την εταιρική νομική ευθύνη. Το δεύτερο είναι ρόλοι και ευθύνες των ενδιαφερομένων κρατών σε διασυνοριακές υποθέσεις. Το τρί, η τρίτη συνιστόσα είναι η υπέρβαση οικονομικών εμποδίων στις νομικές αξιώσεις και απαιτήσει. Το τέταρτο είναι κυρώσεις ποινικού δικαίου. Το πέμπτο είναι ένδικα μέσα ε, με βάση το δίκαιο και το έβδομο είναι η ενίσχυση του έργου των ε, ε, αρχών υπεύθυνων για την εφαρμογή. Έχουμε λοιπόν αυτές τις έξι που είναι σημαντικά διασυνδεδεμένες ε, υπάρχουν διαβουλεύσει με νομικού εμπειρογνώμονε, είτε επειδή υπάρχουν βασικά θέματα που πρέπει να επιληθούν ή να διευκρινιστούν για να υπάρχει συνέχεια και πρόοδος ή γιατί υπάρχει δυνατότητα τα κράτη να κάνουν σαφείς βελτιώσει βράχη και μέσω πρόθεσμα. Το υπόλοιπο της ομιλίας μου θα αναπτύξω περισσότερα θέματα για κάθε συνιστόσα και γιατί κάθε συνιστόσα είναι προτεραιότητα και θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες σε σχέση με τις συνιστώσεις. Ας πάμε τώρα στην πρώτη συνιστόσα του έργου που έχει να κάνει με νομικές ε, δοκιμές για τις καταχρηστικές πρακτικές και την εταιρική νομική ευθύνη, γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλές λεπτές και άλλα και μεγάλες διαφορές στα νομικά κείμενα στις διάφορες δικαιοδοσίες. Αυτό είναι απόλυτα αναμενόμενο γιατί Όλα τα καθιστώτα αστικού και ποινικού δικαίου δεν είναι ακριβώς τα ίδια, ούτε αναμένεται να είναι ακριβώς τα ίδια. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ε, δικαιοδοσίας, ε, όπου μπορεί κάποιος να έχει ευθύνη ε, και βεβαίως διαφέρει και η μέθοδος καταλογισμού. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες διασυνοριακά. Και σε τελευταία ανάλυση κάτω από πανομοιότυπες συνθήκες ε, μια ομάδα θυγωμένων θα έχουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα, μια άλλη ομάδα δεν θα έχει. Άρα αυτό οδηγεί σε ανισότητα σε ό,τι αφορά την νομική προστασία και τα επίπεδα προστασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων και υπάρχει διαφορά γιατί δεν είναι ίση η όρη του παιχνιδιού ε, προκειμένου περί των επιχειρήσεων και εταιριών. Δεύτερη κουκίδα Πολλές φορές τα νομικά καθεστώτα δεν έχουν σαφήνεια σε ό,τι αφορά το πότε θα είναι και πότε δεν θα είναι υπεύθυνη μια εταιρεία. Στην έρευνά μας, και όπως είπε και η Λένε, κάναμε εκτενή έρευνα σε πολλά δικαιικά συστήματα και είδαμε ότι τα νομικά καθεστώτα απλώς δεν είναι ξεκάθαρα σχετικά με τη φύση και το πεδίο εφαρμογής τη εταιρική και αστική ευθύνη. Μπορεί δηλαδή τα νομικά καθεστώτα να μην διευκρινίζουν απόλυτα αν ε, αναφέρονται στις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για τον καταλογισμό ποινικής ιαστικής ευθύνης ή τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ ευθύνης μεταξύ διαφορετικών τμήματων ομίλων εταιριών. Η νομική αβεβαιότης αποτελεί αβεβαιοτηση αποτελει προβλημα και για τις εταιρείες και τα θύματα. Χωρίς τη νομική ασφάλεια ε, όλοι δεν έχουν σαφή βάση για τη λήψη αποφάσεων, για τη νομική ε, ε, δράση, την ε, αντίδραση και αυτό υπονομεύει την ασφάλεια που χρειάζεται για σαφείς επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη σε τελευταία ανάλυση. Τέταρτον, η νομική αβεβαιότητα προσθέτει στο κόστος και το ρίσκο της διαφοράς και της ε, ποινικέ διώξεις. Αυτό είναι πολύ αλήθεια και υπάρχει εδώ μια διασύνδεση με τη συνιστόσα 3 που αφορά τις οικονομικές, ε, τα οικονομικά εμπόδια στις νομικές απαιτήσεις. Θα επανέλθω σε αυτό. Τέλος, ε, υπάρχει έλλειψη σαφών και συνεκτικών δοκιμών για την εταιρική ευθύνη που υπονομεύει την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των νομικών καθεστώτων. Η αποτελεσματικότητα των νομικών καθεστώτων δεν έχει μόνο να κάνει με την δυνατότητα αποτροπής αλλά και τον μηχανισμό ε, αποζημίωσης, τους μηχανισμούς αποζημίωσης και επανόρθωσης. Όπως είπε η Λένε, το σχέδιο αυτό οδηγιών ε, ακολουθεί μια σειρά καλών κρατικών πρακτικών ε, σε σχέση με τέσσερις στόχους κλειδιά Καταρχήν θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η δυνατότητα εταιρική νομικής ευθύνης για εταιρική συμπεριφορά που οδηγεί σε καταχρηστικές πρακτικές. Ε, δεν υπάρχει το τεκμήριο ότι η εταιρική ευθύνη εδώ κατά ανάγκη θα πρέπει να είναι ποινική ευθύνη γιατί σε κάποιες δικαιοδοσίες αυτό δεν αποτελεί δυνατότητα και υπάρχουν πάρα πολλοί νομικοί περίπλοκοι λόγοι γι' αυτό. Αυτός ο στόχος λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει κάποια λογοδοσία νομική, μπορεί να είναι αστική ευθύνη, μπορεί να είναι διοικητική ή ιονή ποινική ευθύνη. δεύτερο δεύτερος πολιτικός στόχος είναι να διασφαλίσει ότι υπάρχει δυνατότητα εταιρικής νομικής ευθύνης σε περιπτώσεις ε, συνενοχής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ε, παράλληλη ευθύνη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ε, σοβαρών καταχρηστικών προακτικών από το στρατό ή την αστυνομία και τέτοια ε, όργανα του κράτους, κρατικούς φορείς. Ε, εδώ μπορεί να μην είναι το κράτος ο βασικός αυτούργος. Θα ανέμενε κανείς να υπάρχει μια σαφής δήλωση στα νομικά καθεστώτα σχετικά με την εισφορά και την εταιρική γνώση και το επίπεδο αυτής που απαιτείται και πώς ε, αυτή αξιοποιείται για να καταλήξουμε σχετικά με την νομική ευθύνη μιας εταιρείας. Όμως τα νομικά πρότυπα και οι κανόνες ε, σπάνια είναι σαφέστατοι και όταν είναι δεν μπορούν να ε, μεταφραστούν πολύ καλά στο εταιρικό πλαίσιο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείε. Ο τρίτος πολιτικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δοκιμές για την ε, νομική ευθύνη των εταιριών ευθυγραμμίζεται καλά με την ανάγκη διαχείρισης κινδύνων από τις εταιρείε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όπου χρειάζονται οι δοκιμές εταιρικής νομικής ευθύνης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που γίνονται από την ε, διεύθυνση να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα ε, ε, τα, τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έγιναν από τις εταιρείε να, να, να αντιμετωπίσουμε τους εργαζομένους ε, υπεύθυνα υπογραμμίζοντας ε, τη λήψη αποφάσεων που γίνεται βάση στιβαρών και αξιόπιστων κανόνων. Υπάρχουν βέβαια πλαίσια όπου για διάφορους πολιτικούς λόγους η αυστηρή, η απόλυτη αυθύνη μπορεί να είναι καλύτερη. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή ε, δεν ε, υπάρχει το θέμα της δέουσας επιμέλειας ή φροντίδας. Και περνάω στην τελευταία δήλωση, πολιτική δήλωση που σκοπό έχει να ε, διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν υψηλά επίπεδα επαγρύπνησης. Γιατί τα εθνικά δικαιικά συστήματα ε, το προβλέπουν, ε, το προβλέπουν αυτό με την έννοια ότι απαλήφουν προσκόμματα ε, σε σχέση με τα ένδικα μέσα και την επανόρθωση όπου αναμένεται ότι μπορεί οι ετούντες να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν την υπόθεση και να στοιχειοθετήσουν την απέτηση αξίωσή τους και σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη χρησιμοποιούν περισσότερο την αυστηρή ευθύνη. Από την άλλη πλευρά, συχνά οι κυρώσεις είναι μικρότερες για να λάβουν υπόψη το μειωμένο επίπεδο ευθύνης και θα επανέλθω στις κυρώσεις σε λίγο. Και τελευταίο σημείο που έχει να κάνει ε, στο τελευταίο, δηλαδή τον, ε, την επίσημη επανεξέταση επανέλεγχο, εμείς ε, θεωρούμε ότι Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση σε κάθε ε, δικαιοδοσία και δικαιικό σύστημα εις ό,τι αφορά την εταιρική νομική ευθύνη. Όμως ο εντοπισμός τομέων υποβελτίωση είναι θέματα που αφορούν την κάθε δικαιοδοσία χωριστά και πολλές φορές χρειάζεται επίσημος ε, νομικός επανέλεγχος ε, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών έχουν ένα μοντέλο, ένα ε, σχέδιο ε, αρμοδιοτήτων το οποίο δημοσιεύεται μαζί με το σχέδιο των οδηγιών. Ε, όμως σίγουρα θα χρειαστούν κάποιες προσαρμογές για να λάβουν υπόψη τα τοπικά δεδομένα. Περνάμε στην επόμενη συνιστόσα, δηλαδή διασυνοριακές περιπτώσεις και ευθύνε των ε, ενδιαφερομένων κρατών. Γιατί αυτό είναι προτεραιότητα, γιατί υπάρχει έλλειψη σαφήνεια ε, σε διεθνέ επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, κατάλληλη χρήση εξοεδαφικής δικαιοδοσία σε διασυνοριακές περιπτώσει. Υπάρχουν προκαταρκτικά έργα που έχουν γίνει για να αποκτήσουμε καλύτερη ιδέα σε σχέση με την στάση και τις στάσεις που υπάρχουν ε, στο θέμα της εξωγραφικής ε, δικαιοδοσίας και για να καταλάβουμε αν υπάρχουν επιμέρους στάσεις που πρέπει να τις γνωρίζουμε. Είναι δύσκολος αυτός ο τομέας γιατί η πρακτική του κράτους μπορεί να είναι αρκετά αυθαίρετη και να εξαρτάται από διάφορα κανονιστικά πλαίσια και οι δηλώσεις των κυβερνήσεων σε σχέση με την χρήση της εξεδαφικής ε, ε, δικαιοδοσίας ε, που πολλές φορές δεν λαμβάνει την υπόψη όπως πρέπει. Βεβαίως υπάρχουν κάποια καθεστώτα που προβλέπουν διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη να αναλάβουν δράση σε σχέση με την εξεδαφικότητα όταν έχουν τη δικαιοδοσία να το κάνουν αυτό. Αλλά πέρα από αυτό το πλαίσιο της συνθήκης οι διατάξεις είναι ακόμα πολύ ασαφείς. Ε, ο δεύτερος λόγος ε, που, ε, γιατί είναι προτεραιότητα αυτό είναι ότι υπάρχει έλλειψη σήμερα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ ενδιαφερομένων κρατών σε θέματα που αφορούν την ανείχνευση, τον εντοπισμό, την έρευνα, την δίωξη και την επιβολή. Εδώ υπάρχουν πολλά διεθνή καθεστώτα τα οποία προβλέπουν συνεργασία διακρατικά ε, όταν πρόκειται για την έρευνα και την δίωξη κρεπινικών δραστηριοτήτων και υπάρχουν και καθεστώτα που προβλέπουν μηχανισμούς όπου η νομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί και να παρασχεθεί και σε αστικές υποθέσεις. Όμως οι εισαγγελίες μας λέγουν ότι η εφαρμογή πολλές φορές δεν είναι καλή και στην πράξη υπάρχουν πρακτικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, προβλήματα επικοινωνίας που επηρεάζουν αρνητικά την συνδρομή. Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και συντονισμού επίσης και ακριβώς γι' αυτό είναι προτεραιότητα αυτό το θέμα για μας. Όλα αυτά δημιουργούν νομική ανασφάλεια, ε, εμποδίζουν την ικανότητα των εισαγγελέων να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες, ανεβάζουν το κόστος και την συνθετότητα των υποθέσεων και υπονομεύονται οι προσπάθειες των εθνιστικών φορέων να προλάβουν, ανοιχνεύσουν και να ε, ε, επιβάλλουν τον νόμο σε διασυνοριακές υποθέσεις. Και πάλι λοιπόν η οδηγία αυτή ο προσανατολισμός λαμβάνει υπόψη μια σειρά καλών κρατικών πρακτικών με βάση ε, έξι πολιτικούς στόχους. Τα κράτη θα πρέπει να κατανοήσουν όσο γίνεται πληρέστερα τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνή και εθνικά καθεστώτα αυτή τη στιγμή ε, λύνουν διασυνοριακά προβλήματα και τι δυνατότητα έχουν να αναπτυχθούν στο μέλλον και οι πολιτικοί αυτοί στόχοι έχουν να κάνουν με την διευκρίνηση από τα ίδια τα κράτη των διαφορετικών πλαισίων όπου η εξεδαφικότητα και η μέθοδοι της μπορεί να είναι υποφελής και εκεί όπου μπορεί να απαιτούνται στα πλαίσια διεθνών καθεστώτων. Ο δεύτερος στόχος είναι να μπορέσουν η ε, δικαστική εξουσία να ζητήσει συνδρομή άλλων δικαιοδοσιών. Τα στοιχεία καλής ε, ορθής πρακτικής ε, στοιχειοθετούν διαφόρους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική διεθνή συνεργασία τα κράτη και να διασφαλίσουν ότι οι σωστές διευθετήσεις υπάρχουν ρυθμίσεις σε νομικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο και βεβαίως οι δικαστικοί θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, υποστήριξη και ε, θα πρέπει να υπάρχουν και κοινέ ομάδες έρευνας. Αυτές απεδείχθησαν ότι είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνιστούν ένα μοντέλο που αρχίζει να βρίσκει μιμητές και αλλού. Ο τρίτος πολιτικός στόχος είναι πολύ πρακτικός, αφορά την Συμφωνία σε κοινέ προσεγγίσεις για την βελτίωση και επιτάχυνση της ε, συνεργασίας. Θα πρέπει να υπάρχουν δηλαδή κοινέ νόρμες ε, και διαδικασίες ούτω ώστε να διευκολύνονται οι επαφές, ε, η πρόσβαση σε πληροφορίε, οι έρευνες και να μπορούν οι εισαγγελίε και οι δικαστικοί, οι νομικοί να διευκολύνεται στο έργο τους. Και υπάρχουν και άλλοι δύο πολιτικοί στόχοι που έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ε, καλύτερης πρόσβασης στις συνοριακές πληροφορίες και σταδιακή βελτίωση των καθεστώτων, τόσο ώστε να ενισχύουν, να εμβαθύνουν τη συνεργασία και περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Τώρα, υπέρβαση οικονομικών εμποδίων. Ε, και αυτό έχει να κάνει με την τρίτη συνιστόσα. Εδώ έχουμε μία προτεραιότητα ε, για ένα θεμελιώδη λόγο. Άνθρωποι που επηρεάζονται αρνητικά. Ε, εδώ Πολλές φορές έχουν μεγάλο πρόβλημα ε, με τα ένδικα μέσα και την επανόρθωση. Αυτό βεβαίως υπάρχει σε, όλες τις, ε, ε, όλα τα δικαιικά συστήματα. Εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχουν διαφορές. Πολλές φορές αυτό οφείλεται σε ευρύτερες προκλήσεις, νομικές και οικονομικές επίσης. Μία από αυτές τις προκλήσεις έχει να κάνει με την συρρήκνωση των κρατικών προϋπολογισμών για την νομική διαρρογή που αυτό είναι μια σαφή τάση και η ομάδα μας βεβαίως ήθελε να δει και τι άλλες πηγές χρηματοδότησης μπορούν να εξεταστούν και να χρησιμοποιηθούν σε όλο τον κόσμο. Εδώ συλλέγουμε ακόμα στοιχεία. Αλλά όταν μιλάμε για οικονομικά εμπόδια υπάρχουν δύο σκέλη στην εξίσωση. Υπάρχει η δυσκολία να βρεθεί χρηματοδότηση και υπάρχει και το άλλο σκέλος. Υπάρχει και η πλευρά του κόστους των δαπανών τα δικαστικά έξοδα είναι πολύ υψηλά πολλές φορές. Βλέπουμε λοιπόν και τα δύο σκέλη της εξίσωσης και ζητούμε από τους εμπλεκομένους να παρουσιάσουν τρόπους ε, βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Πρέπει επίσης να δούμε και το θέμα της κλιμάκωσης αυτής, της αύξησης των δικαστικών εξόδων και πώς αυτά μπορούν να μπουν υπό έλεγχο. Τώρα, οι βασικές συστάσεις παρουσιάζονται σε αυτήν εδώ την διαφάνεια. Ε, στοιχεία ορθής πρακτικής που αφορούν ε, πηγές χρηματοδότησης, ε, νομική βοήθεια, κρατική, βελτίωση στη χρηματοδότηση από, τα, από τους διαδίκους, τους ασφαλιστές, ε, ρυθμίσεις ε, σχετικά με έκτακτες αμοιβέ, συλλογικές δράσεις και δυνατότητες τέτοιας διαχείρισης ε, που μεταξύ άλλων θα μειώνει το, τα έξοδα και θα ε, δίνει ε, κίνητρο για καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα, προσβασιμότητα και αποτελεσματικότητα. Τώρα, η τέταρτη συνιστόσα, ποινικέ διοικητικέ κυρώσεις και αυτό είναι προτεραιότητα γιατί διότι στην πράξη η εφαρμογή και η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε εταιρείε ε, όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα είναι σπάνιες, ε, μπορούν καμιά φορά να ε, ισχύσουν και σε πολίτες, σε μονομένα πρόσωπα, αλλά δεν έχουμε ερευνήσει αρκετά το θέμα των εταιρικών ποινικών κυρώσεων που μπορεί να εφαρμοστούν θέλουμε να δούμε εάν είναι αποτελεσματικές. Στην πράξη και προς το παρόν οι ποινικέ εταιρικέ ε, κυρώσεις ε, πολλές φορές ε, δεν δρούν αποτρεπτικά, δεν διασφαλίζουν την μία επανάληψη της ζημίας, δεν είναι αποτελεσματικός αποζημιωτικός μηχανισμός. Εδώ δεν είδαμε μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, πήραμε και παραδείγματα από άλλα εθνικά δικαιικά συστήματα που ε, αφορούν θέματα ε, ε, καταπολέμησης διαφθοράς, προστασίας περιβάλλοντος, πλαίσια της εταιρικής ευθύνης. Και όπως βλέπετε εδώ τα στοιχεία καλής πρακτικής εδώ καλύπτουν θέματα όπως αποτροπή, ε, τι πράγματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζουμε τις κυρώσεις, συμπεριλαμβάνοντας οικονομικές κυρώσεις, τη δυνατότητα αποζημίωσης. Είναι σημαντική η ανάγκη σωστής διαβούλευσης με τα θύματα για να εξετάσουμε και τα προγράμματα συμμόρφωσης των εταιριών, ε, δέουσα επιμέλεια, δέουσα φροντίδα κλπ. Πέμπτη συνιστόσα. Ε, αυτή είναι προτεραιότητα γιατί τα ένδικα μέσα αστικού δικαίου στην πράξη σπάνια πληρούν τα διεθνή πρότυπα ε, της κατάλληλης αποτελεσματικής άμεσης ε, ε, αποζημίωσης και επανόρθωσης. Και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των δικαιικών συστημάτων σε ό,τι αφορά τα ένδικα μέσα στο αστικό δίκαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Ε, έτσι δημιουργούνται ενισότητες μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω έλλειψης διαβουλεύσεων με τις ομάδες ενδιαφερόντων και κοινότητες σε ό,τι αφορά το τύπο του ένδικου μέσου που απαιτείται. Έτσι υπάρχει αναποτελεσματικότητα και υπάρχει και έλλειψη σαφήνειας σε ό,τι αφορά τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να διέπουν την κατανομή των ζημιών στις ομαδικές απαιτήσει αξιώσεις, δηλαδή πώς καθορίζουμε ε, τα πρόσωπα που θα αποζημιωθούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν πρόκειται για κατανομή ε, μεταξύ ομάδων ε, περιθωριοποιημένων ή ευπαθών ετούντων. η απάντηση του οδηγού ε, με τις, ε, είναι ε, μια απαρίθμηση ορθών πρακτικών από την έρευνα που λαμβάνει υπόψη θέματα όπως μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η ζημία, εναλλακτικέ σε οικονομικές αποζημιώσεις, ανάγκη για διαβουλεύσεις με τα θυγόμενα πρόσωπα, στην περίπτωση διακανονισμού διαβουλεύσεις με τους θυγωμένους σε ό,τι αφορά τους όρους του διακανονισμού και η ανάγκη να υπάρχουν κάποια πρότυπα για την δίκαιη κατανομή των ε, εσόδων, των, αποζημιώσεων ε, όταν είναι ομαδικές οι απαιτήσει. Τέλος, ε, εις ό,τι αφορά την δίωξη και επιβολή του νόμου, και αυτό είναι προτεραιότητα για μας, γιατί τα επίπεδα δραστηριότητας από τις διοκτικές αρχές σε ποινικά θέματα ε, είναι πολύ ε, χαμηλά σε περίπτωση ε, εταιρική συμμετοχή σε σοβαρέ καταχρηστικέ πρακτικέ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε όμω υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητα σε πιο κωδικοποιημένου τομεί, για παράδειγμα εργατικό δίκαιο, περιβαλλοντικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντο. Ε, και έχουμε συζητήσει με εισαγγελίες, έχουμε μιλήσει και με τη Διεθνή ε, Αμνηστία και έχουμε συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις και στρογγυλά τραπέζια πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, και χωριστά επίσης πήραμε πολλές συνεντεύξεις από εισαγγελίες σε πολλές, από πολλές χώρες και συζητήσαμε και με τη Διεθνή Ένωση των Εισαγγελέων Αυτέ ε, τα αποτελέσματα αυτών των ε, συζητήσεων και συνεντεύξεων ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ανέδειξαν πολλά προβλήματα που πρέπει να ε, εξετάσουμε για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της Επιβολή του νόμου, υπάρχει έλλειψη, όπως είδαμε, κατάρτισης πόρων, πρακτικές δυσκολίε που αφορούν τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, προβλήματα σε σχέση με τον εκφοβισμό των μαρτύρων, ε, επίση ε, ε, νομικές πολυπλοκότητες και έλλειψη πολιτικής και διοικητικής υποστήριξης. Οι συστάσεις λοιπόν που αφορούν ορθές πρακτικές περιλαμβάνουν ε, την ανάγκη ε, για για πολιτική και δικητική υποστήριξη, αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των κρατικών ε, αρχών και φορέων. Υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων που αφορούν την διακριτική ευχέρεια των εισαγγελικών και διοκτικών αρχών και διάφορες προτάσεις που αφορούν την εκπαίδευση, τους πόρους, την τεχνογνωσία, την πραγματογνωμοσύνη, πώς δημιουργούνται ικανότητες σε διασυνοριακές υποθέσεις, προστασία μαρτύρων και τέλος τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται ε, σε επίπεδο επαγγελματισμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού από τις ε, βιοπτικές ε, και εισαγγελικές αρχές. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε ερωτήματα. Ε, ναι και ένα μικρό σχόλιο. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο μιλήτριες ε, για ε, την παρουσίασή τους πάνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ε, κάνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και, για πιο, ε, και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι γίνεται στο πλαίσιο της Ολλανδικής ε, Προεδρίας η οποία έχει θέση ε, την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά ως έναν από τους βασικούς της τομείς, ενώ επιπρόσθετα η Κομισιόν ε, προετοιμάζει ένα σχέδιο Α δράσης ε, σχετικά με την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά. Δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς είναι ο τίτλος του, όμως πιστεύω ότι μια ομάδα επιτρόπων θα εξετάσει όλη αυτή την περιοχή που είναι ιδιαίτερα μεγάλη και σύμφωνα με τις πηγές που έχω από την Κομισιόν ε, το ε, πρώτο προσχέδιο θα υπάρχει ε, κατά το Μάιο φέτος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Επιπλέον στο Κοινοβούλιο ε, μπορώ να υπολογίσω ότι υπάρχουν 5-6 επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων είναι επιτροπή που συνδέεται άμεσα με το ε, ζήτημα των επανορθώσεων Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να, μπορέσουμε, θα μπορέσουμε να βρούμε το πού ταιριάζουμε εμείς σε αυτό το έργο. Τώρα το ερώτημά μου προς τις ε, ομιλήτριες είναι πώς περιμένετε ένας τέτοιος υπερεθνικός οργανισμός όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει ε, να συμμετάσχει και βέβαια το έργο σας ακόμα εξελίσσεται, όμως παρόλα αυτά έχουμε δει σημεία κλειδιά. Ποιε λοιπόν είναι οι συνέπειες ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος του ήθελε επίσης να θέσει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ. Η προσπάθεια την οποία κάνει η υπηρεσία της ΥΠΑ της Αρμοστίας είναι ιδιαίτερα προχωρημένη. Προκαλεί ενδιαφέρον το θέμα και στην ουσία η προσπάθεια αυτή τη μάθα, ε, έλεγα ε, τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες αυτές έρευνες. Δεν είναι τυχαίο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα πέρυσι και ακόμα πιο πρόσφατα συγκέντρωσε την προσοχή του στον ρόλο τον οποίο μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της λεγόμενης θετικής διακυβέρνησης. Και έχουμε μαζί με το θέμα της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης Έχουμε επίσης συζητήσει και το θέμα των μη οικονομικών επανορθώσεων. Ο λόγος είναι γιατί όχι μόνο θα πρέπει να ενισχύσουμε τις θετικές πλευρές οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στο εσωτερικό της αποστολής της επιχείρησης αλλά να εντοπίσουμε και σαν μια επιπλέον υποχρέωση για τις επιχειρήσεις το θέμα της αναγνώρισης των ευθυνών όχι μόνο για αυτά τα οποία κάνει η επιχείρηση αλλά και για αυτά τα οποία επιβάλλει οι άλλοι να κάνουν στις διαδικασίες τις υπεργολαβικές είναι σαφές από ορισμένε επιχειρήσεις να δίδουν σε άλλους υπεργολάβους το πιο επικίνδυνο και αρνητικό τμήμα των αρμοδιοτήτων τους, να εκχωρούν αυτές τις επικίνδυνες λειτουργίες. Οπότε η ευθύνη για πιθανές κυρώσεις ε, σε συγκεκριμένες τέτοιες δράσεις Στα πλαίσια της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις η ανάληψη της ευθύνης είναι σαφής. Πρώτον θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε κάποια ποσοτικά στοιχεία για τις αρνητικές συμπεριφορές στα πλαίσια των υπεργολαβιών. Ξέρω ότι εδώ ισχύει περισσότερο εθνικός κανονισμός και δεν υπάρχει ομοφωνία θέλετε και ενιαία εικόνα σε κάθε χώρα. Δεύτερον, πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο και εγώ το πιστεύω αυτό να εφαρμόσουμε αυτά που είχαμε ψηφίσει πρόσφατα σε σχέση με την ευθύνη των επιχειρήσεων και τις μη οικονομικές επανορθώσεις. Δηλαδή στα πλαίσια της διακυβέρνησης ε, του θέματος γενικότερα της επιχειρηματικής ευθύνης θα πρέπει θα έλεγα το στοιχείο αυτό να καταστήσει σημείο ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συμβαλωμένων γενικά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει ε, μια κανονική υγιής, θα έλεγα, συμπεριφορά από πλευράς μιας επιχείρησης ή ενός υπεργολάβου, θα πρέπει να τίθεται το θέμα της ανάληψης της ευθύνης και των συνεπειών της. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά το γεγονός ότι ξεκινούμε μια νέα ψηφιακή ε, περίοδο όπου ιδιαίτερο στα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική σφαίρα δέχεται έντονη πίεση. Υπάρχουν λοιπόν δεδομένα πάνω σε αυτό το ζήτημα και ε, δεύτερον όπως είπε η συνάδελφος Χάουτελε, αν έχουν βγει κάποιες ε, υποχρεώσεις, ε, θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν έχει, έχετε ε, βρει κάποια ελλείμματα στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κράτη-μέλη της, Ιδιαιτέρως μάλιστα θα έλεγα διότι τα τελευταία χρόνια εφαρμόσαμε νομοθεσίας που αφορούσαν την προστασία θυμάτων και θα έλεγα ε, κατά πόσο αυτά συμφωνούν ε, με το δικό σας έργο. Εσείς θα, εσείς θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε εντοπίσει κάποια ελλείμματα πάνω σε αυτό. Ωραία, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ε, θα, θα μπορούσατε να δώσετε σύντομες απαντήσεις διότι μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τα ερωτήματα. Ε, χαιρετίζω ιδιαίτερως ε, το γεγονός ότι η Ολλανδική ε, Προεδρία επικεντρώνεται πάνω στην εφαρμογή των κατευθυντήριων του ΟΗΕ και αδειμονούμε να δούμε και το σχέδιο δράσης της Κομισιόν ε, δεν ξέρω αν θα επικεντρωθεί στην ε, στάση των ε, επιχειρήσεων και αν συμφωνεί απόλυτα με το δικό μας έργο, όμως παρόλα αυτά το χαιρετίζουμε και θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα όσον αφορά τα ζητήματα ε, της επικέντρωσης ε, του, του ζητήματος πάνω στο οποίο θα επικεντρωθεί η ίδια η ε, Προεδρία της Ολλανδίας η οποία δεν θα επικεντρωθεί μονάχα στο έργο λογοδοσίας και επανόρθωσης αλλά θα αναφερθεί και σε ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν από τους διάφορους ομιλητές. Νομίζω αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία Τώρα όσον αφορά ένα υπερεθνικό σώμα όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία κατευθυντηρίων αλλά και τη χρήση των κατευθυντηρίων ούτως ώστε να ενσωματεθούν στη συνέχεια σε, οδηγίε οδηγίες αλλά και σε άλλες πολιτικές Επίσης όσον αφορά την ε, διακυβερνητική ομάδα του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διακυβερνητική συνεργασία, το έργο λογοδοσίας ε, και ε, επανορθώσεων είναι ουδέτερο και οι προτάσεις μπορούν να υιοθετηθούν από εθνικές κυβερνήσεις που προσπαθούν να βελτιώσουν το νομικό του σύστημα σύστημα, όμως ε, ταυτόχρονα μπορεί να υιοθετηθεί και στο σύνολο από διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν όσον αφορά το, το γεγονός ότι βασιζόμαστε ε, σε συγκεκριμένες εντολές ε, διεθνώς οργανισμών και περιφερειακών οργανισμών, Νομίζω ότι οποιαδήποτε εντολή η οποία σχετίζεται με τις επανορθώσεις που αφορούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και να υιοθετήσουμε πολλά και γι' αυτό το λόγο έχουμε ε, και πολυμερείς θεσμούς ούτω ώστε ε, να έχουμε και υπερεθνικές ε, νομοθεσίες και να δοθούν κατευθυντήριες σχετικά με το πώς θα πρέπει να είναι οι οδηγίες αυτές. Γι' αυτό το λόγο καλώ την Επιτροπή αυτή και άλλες επιτροπές τις οποίες αναφέρατε, οι οποίες ίσως να σχετίζονται με το θέμα αυτό, να ελέγξουν τις κατευθυντήριες τις οποίες θα δημοσιεύσουν, ευσιεύσουμε και να δουν πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ε, πάνω ε, στο έργο σας. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα των ε, παρόχων και των ποσοτικών δεδομένων, Πολύ συχνά όταν μιλούμε για το πρόγραμμά μας λέμε ότι είναι ένα ε, πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ ε, μεγάλο σκοπό και αφορά μια σειρά νομοθετικών ε, ζητημάτων. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένει ταπεινό διότι παραμένει στα έξι σημεία τα οποία στα οποία επικεντρωνόμαστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία μπορούν να συσχετιστούν όπως είναι η διαφορά η εφαρμογή των κατευθυντηριών του ΟΗΕ όσον αφορά την παροχή ε, υπηρεσιών. Είναι ζητήματα στα οποία επίση ασχολούμαστε. Όλα αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία έχουμε ελέγξει αναλυτικά στο πλαίσιο του έργου μας διότι προσπαθήσαμε να παραμείνουμε συγκεκριμένοι πάνω στα ζητήματα στα οποία θέλαμε να επιτύχουμε πρόοδο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα όμως ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα διαδικαστικά ζητήματα όσον αφορά ε, τα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία ε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ε, έρευνα του δικού μας προγράμματος. Σε άλλα μέρη λοιπόν του έργου μας, όπως ανέφερα, Υπάρχουν ε, πάρα πολλές σημαντικές ε, αναφορές ε, σχετικά με το έργο αυτό και γίνονται σε διάφορους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε το έργο των εταιριών όταν το ζήτημα αφορά τα, τον κίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αλυσίδα ανεφοδιασμού. Παρομοίως όσον αφορά την ε, ψηφιακή εποχή, Πρόκειται και πάλι για ένα ζήτημα το οποίο αφορά ιδιαίτερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει συζητηθεί ιδιαίτερο στο πλαίσιο του ε, Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από τον ε, το αρμοστή σχετικά με την ε, ελευθερία έκφρασης. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στον ψηφιακό τομέα ο Ήπατος ε, αρμοστής την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα έδωσε μια ε, ανακοίνωση σχετικά με τη διαμάχη μεταξύ της Apple και του FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως εγώ θα περιοριστώ στο δικό μου έργο Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα πάρα πολύ να σας παραπέμψω σε αυτούς οι οποίοι είναι ε, πιο ε, καλά καταρτισμένοι σχετικά με αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα τα ελλείμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Έχουμε ε, πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς θα είναι αυτό, όμως για το σκοπό αυτού του έργου, έργου δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε στις συγκεκριμένες χώρες και να αναφέρουμε συγκεκριμένες χώρες, για τον σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος. Υπάρχει ένα αμάλγαμα των δεδομένων τα οποία έχουμε, το οποίο να μην περιλαμβάνει μια τακτική όπου ονομάζουμε και ντροπιάζουμε, αλλά είναι μια τακτική όπου θα έχουμε, αλλά σε μια διαφορετική φάση αυτού του προγράμματος θα εξετάσουμε αν μπορέσουμε να λάβουμε εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το πώς θα ανταποκριθεί πάνω σε αυτό και στη συνέχεια ε, θα κάνουμε μια ε, περαιτέρω έρευνα σχετικά με, το, ε, με τα κράτη-μέλη, το, πώς το πώς θα πηγαίνουν πάνω σε αυτό και το πώς προωθούμε πρακτικές και το πώς εφαρμόζονται όμως για την ώρα θα επικεντρωθούμε σε μια πιο γενική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ε, ελπίζω λοιπόν τα μέλη να έχουν λάβει τις αναγκαίες απαντήσεις. Ε, φαίνεται πως έτσι έχει κατάσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κυρίες μου που ε, βρισκόσασταν σήμερα μαζί μας και μας δώσατε ε, πληροφορίες για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, ε, το οποίο αφορά την ανταλλαγή από, ε, απόψεων σχετικά με την ευθύνη αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και φυσικού αερίου και πριν δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή κύριο Χρυσόγωνο θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Στέφαν Μόζερ και τον κύριο Γιάνν Λάμπη, οι οποίοι οι οποίοι θα δώσουν αναφορά, οι οποίοι θα σχολιάσουν τη συγκεκριμένη αναφορά. Θα ήθελα όμως αρχικά να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν ε, την ε, εταιρική ευθύνη όσον αφορά την, ε, ε, την ε, έρευνα και την εξόριξη πετρελαίου. Μέχρι στιγμής η Ευρώπη δεν έχει αντιμετωπίσει ατυχήματα όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβη τον Απρίλιο του 2010 στην εξέδρα Deep Horizon στον κόλπο του Μεξικού. Η σοβαρότητα τέτοιων ατυχημάτων και των συνεπειών τους δικαιολογεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, προβλέψεις για αυτό. Το 73% ε, της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αέριου προέρχεται από ε, κράτη-μέλη της Βόρειας Θάλασσας που ήδη εφαρμόζουν τα πιο αυστηρά καθεστώτα ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η εναρμόνιση του νομοθετικού, πλαισίου, νομοθετικού δεν είναι κάτι για αυτές τις χώρες. Όμως ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια μεγαλύτερη παραγωγή και εξόρυξη πετρελαίου από άλλα κράτη-μέλη επίσης, όπως είναι για παράδειγμα η Κύπρος, όπου υπάρχουν μεγάλα αποθέματα, παράκτια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και γι' αυτό το λόγο το νομοθετικό πλαίσιο της οδηγίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας καθότι επιβάλλει την διάβγεια και ε, καθιστά την αναγκαιότητα ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά ατυχήματα και παρολίγων ατυχήματα, καθώς επίσης ε, και δείκτες αποδοτικότητας ε, στον τομέα όσον αφορά την ασφάλεια. Η αναφορά της Κομοσιόν αφορά διάφορα ζητήματα όπως είναι, όπως είναι η επιχειρηματική υπευθυνότητα, όπως για παράδειγμα ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί ατύχημα και γιατί απώλειος απέναντι σε ποιον ενώ το άλλο ζήτημα αφορά ότι ε, τα ε, συμπληκόμενα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ε, την επαρκή αποζημίωση για την βλάβη που προκάλεψαν. Ενώ τρίτον, ποιος είναι ο τρόπος για την αποζημίωση και το πώς αυτός η αποζημίωση αυτή θα μπορέσει να δοθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα θύματα. Η Κομισιόν δηλώνει τέλος ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες επανορθώσεων ε, αποδίδουν δικαιοσύνη στα θύματα τέτοιων ατυχημάτων. ατυχημάτων. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν λέει ότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι προσεγγίσεις αυτές είναι λιγότερο αποτελεσματικές όσον αφορά την ασφάλεια των υπεράκτιων ε, δραστηριοτήτων εξόριξης. Η Κομισιόν λοιπόν δηλώνει ότι η εφαρμογή της οδηγίας στον, στην εθνική νομοθεσία θα πρέπει θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2015 συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη να υπάρχει άμεση ε, προσαρμογή της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, όμως ε, δεν συμφωνώ με το συμπέρασμα της Κομισιόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν ποινικέ κυρώσεις ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ε, την υπεράκτη ασφάλεια. Πιστεύω ότι η αποτροπή είναι καλύτερη από τη θεραπεία και η εφαρμογή ποινικών κυρώσεων τώρα θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε τις εναλλακτικέ σε ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την οικονομική ασφάλεια και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια άμεση διαχείριση των ετοιμάτων για αποζημιώσει. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω μιας νέας πράξης ή μέσω τη τροπο, ε, της τροποποίησης της υπάρχουσας, κάτι το οποίο θα είναι πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ε, λάθος ε, οικονομικά μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μόζερ, αν το επιθυμείτε. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που έκανε την παρουσίασή του. Θα συμφωνήσουμε για τη σημασία που έχει αυτό το θέμα και αναγνωρίζουμε το θέμα της ευθύνης έτσι όπως τίθεται και στην έκθεση. Εμείς σαν Επιτροπή πρέπει να ελέγξουμε την εφαρμογή της συγκεκριμένης ε, διάταξης στην εθνική τους νομοθεσία, να δούμε αν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο. Η αξιολόγηση την οποία κάνουμε συνεχίζεται. Πρώτα θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης και όταν το κάνουμε αυτό, τότε θα κάνουμε μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και κάποιες αλλαγές στο πλαίσιο είτε μέσω της τροπολόγησης της οδηγίας είτε μέσω της δημιουργίας ενός διαφορετικού μέσου. Δεν το έχουμε κατορθώσει ακόμα αυτό, βρισκόμαστε στο μέσον της διαδικασίας ελέγχου στα κράτη-μέλη. Μετά θα πρέπει να τα αναλύσουμε αυτά τα οποία θα βρούμε, τα ευρήματα Πάντως η πρόταση για να γίνει συζήτηση στην παρόουσα φάση και τους εμπλεκομένους είναι μια θετική πρόταση να δούμε τι χρειάζονται και οι επιχειρήσεις και επί αυτής της βάσεως θα επανέλθουμε με πιθανές προτάσεις. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Λάμπη. Κύριε Λάμπη θέλετε το λόγο. Όχι, ο κύριος Λάμπη δεν θέλει το λόγο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Άντερσον έχει να κάνει μια ερώτηση. Δεν νομίζω, Πρόεδρε, ότι είναι ερώτηση. Περισσότερο μια γενική παρατήρηση. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την σημαντική συζήτηση. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει. Η ομάδα των πρασίνων δεν είναι και τόσο πρόθυμη όσο άλλοι να συνεχιστούν και να υπάρξουν και νέες μορφές εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Γνωρίζουμε πόσο επηρεάζει το κλίμα αυτό όπως επίσης και το πετρέλαιο. Έχει σημασία πάντως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ε, καταστροφές όπως αυτό το Deep Water, η πλατφόρμα της BP. και να μην χάνονται ποσότητες πετρελαίου που χύνονται στους ωκεανούς. Απαιτούνται σκληροί κανόνες, αυστηροί κανόνες, απαιτούνται κίνητρα για περαιτέρω μορφές συνεργασίας. Και θα πρέπει να γίνει κάθε ε, προσπάθεια αποφυγής ατυχημάτων. Οι διαδικασίες αυτές χρειάζεται να είναι διαφανείς ε, πρέπει να είναι διαφανείς και οι οικονομικές δομές των ε, ασφαλιστικών μέτρων, των μέτρων ασφαλείας μάλλον και ε, των αποζημιώσεων και θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε και τα προβλήματα ηθικού κινδύνου τα οποία μπορεί να τεθούν σε περίπτωση πληρωμών από ασφαλιστικές εταιρείες. Λοιπόν, προσβλέπω με ενδιαφέρον την συνέχιση της προσπάθειας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο από τα διάφορα μέλη. Όχι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο στις παρατηρήσεις του κυρίου Άντερσον. Σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Θα συμφωνήσουμε λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για την ανάγκη να υπάρξει ένα πλαίσιο αποτροπής των ατυχημάτων, ένα πλαίσιο διαφανές και ξεκάθαρο. Όταν διαπραγματευτήκαμε για πρώτη φορά στα πλαίσια της οδηγίας την πρόταση αυτή, εντοπίσαμε και τη βάση στην οποία ακριβώς χρησιμοποιεί και η έκθεσή σας. Το κάναμε με βάση τις γνώσεις τις οποίες είχαμε και στην παρούσα φάση δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το βέλτιστο καθεστώς. Θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα όταν μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την εφαρμογή των μέτρων από πλευρά των κρατών μελών και συγκρίνουμε τα διαφορετικά καθεστώτα. Και τότε θα δούμε τι περαιτέρω μέτρα απαιτούνται. Αυτό θα πρέπει να γίνει μάλλον το 2019 όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. provisions of the Directive are about um, preventing these Πράγματι, στόχος μας είναι η πρόληψη καταστροφικών συμβάντων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της οδηγίας, έτσι όπως καλείται να εφαρμοστεί και στα πλαίσια ε, των αποζημιώσεων και των ασφαλιών. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία τίθενται σε εφαρμογή με στόχο την πρόληψη. Αυτή στιγμή λοιπόν εμείς έχουμε μια σαφέστερη εμπειρία των προληπτικών μέτρων τα οποία εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες μέσω της οδηγίας, τότε θα αξιολογήσουμε καλύτερα το καθεστώς αποζημιώσεων που ισχύει και αυτό προβλέπεται μάλλον να ολοκληρωθεί σαν διαδικασία τον μήνα Ιούλιο του 2019. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλώς. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να έχει ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, ήταν μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ που ήσασταν όλοι παρόντες. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή αυτή. Και κλείνουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο λοιπόν.